So, let me start meeting of our uh, Ξεκινώ λοιπόν τη συνεδρίαση. Θα χρειαστεί να αναγνώσω διάφορα έγγραφα ξεκινώντας πριν περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα λοιπόν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω προτάσεις για τροποποίηση. Ας περάσω στο δεύτερο θέμα που θα μας κρατήσει λίγο περισσότερο. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου της έχει ετοιμάσει η Γραμματεία. Η πρώτη συνεδρίαση της EconFam, 21 ε, Νοεμβρίου. Έχετε ενημερωθεί για την κοινή συνεδρία Τετάρτη το πρωί με ψηφοφορία για την έκθεση πρωτοβουλίας για το, την σωματοστέση του φίλου στις ε, εκθέσει για φορολογικά ζητήματα. Για να μην έχουμε προβλήματα σχέση με τη διεξαγωγή της ε, Tax 3, 3 την ίδια ώρα. Παρακαλώ να έρθετε νωρίς για να προχωρήσουμε. Επίσης, σύνοψη και προτάσεις των συντονιστών, τελευταία συνεδρίαση και διορισμοί 2017 απαλλαγή η ΕΒΑ, ΕΟΠΑ και ΕΣΜΑ ΣΕΝΤΗ Brexit ενημέρωσε ο Πρόεδρος για τις, εξελίξει, για, για τις νέες εξελίξεις, αλλά εντωμεταξύ μας έχει ξεπεράσει η επικαιρότητα. Χρονοδιάγραμμα για την άτυπη ακρόαση της 21 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε, αυτό το μεταξύ έχει διεξαχθεί. Ομάδα εργασίας, α όχι, χρηματοοικονομικής βοήθειας και εποπτεία για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι η ενισχυμένη εποπτεία θα λαμβάνει χώρα στην ΕΚΟΝ και θα συνεχιστεί η δυσχετική δουλειά. Συντονιστές επίσης, προσεχή του συνεδρίες. 10 Οκτωβρίου επίσης έχει διεξαχθεί και στην εν λόγω συνεδρίαση συντάχθηκε το κείμενο για το Μάρτιο για, το επόμενο, για τον επόμενο χρόνο 21 Ιανουαρίου, 26 Απριλίου, 18 Μαρτίου, το γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι οπωσδήποτε, συστάσεις για τον κανονισμό για την ΕΣΑΣ, τροποποίηση της πρότασης επιτροπής, ανταλλαγή απόψεων όπου αποφασίστηκε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Να διατηρηθεί μία έκθεση τροπολογίες. Με ένα μόνο τμήμα. Κατά τη στιγμή των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο θα εξεταστεί αν υπάρχουν ανάγκε για περαιτέρω. Επίση, οικονομικέ εξελίξει. Eurogroup στη Βιέννη 17 Σεπτεμβρίου, όπου αποφασίστηκε εν ώψη προσεχών συνεδριάσεων θα προσκαλείται ο Πρόεδρος και θα προστίθεται το σχετικό θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη για τους τονιστές αμέσως μετά. Επίσης, ε, ομάδα εργασίας για την οικονομική βοήθεια, ενσωμάτωση των θεμάτων, των προτάσεων και πρόταση προς τους ενδιαφερομένους για τη συνεδρία του 2019. Επιτροπή για τον επόμενο χρόνο και χρονοδιάγραμμα έχουμε στην Deutsche Bank μια επίσκεψη τη Δευτέρα της Ολομέλειας στην Deutsche Bundesbank έχει μια διαφορά 28 Φεβρουαρίου επίσης μια επίσκεψη στο Λονδίνο 29 Φεβρουαρίου και 1η, 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου Επίσης, στο σχέδιο μίλησε διάταξη τα σχετικά θέματα θα συμπεριληφθούν στην προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών. Fiscal Compact, γνωμοδότηση της Γιούρη θα ζητηθεί για τις προτινόμενες αλλαγές στην νομική βάση, διάφορα. Αποφασίστηκε κατόπιν ετήματος του αρμόδιου Υπουργού να γίνει ακρόαση για την ψηφιακή φορολογία στις 23 Οκτωβρίου, Τρίτη. Συντονιστές 21 προσεχή συνεδρία των Στον 21 Νοεμβρίου. Μάλλον αυτά είναι όλα από τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Τώρα έχουμε την έκθεση για τις συνεχιζόμενες διοργανικές συνομιλίες, τριμερής διάλογος για ένα BEPS, Πανευρωπαϊκό Σύστημα Συνταξιοδότηση. 15 Νοεμβρίου πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή παρουσίασε τέσσερα non-paper για την ε, ε, μετατροπή, περιεχόμενο, μεταφορετικότητα, μετατροπή, αποθετήρια. 4 Δεκεμβρίου προσοχή συνεδρίαση και έτσι πάμε στο πρώτο μας θέμα και το σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη, αγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματο ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Φούλβιο Ματουσέλο. 25 λεπτά έχουμε στη θέσή μα για τη συζήτηση, αλλά καθώ ο κύριο Μαρτουσέλο δεν είναι εδώ, θα τον εκπροσωπήσει ο κύριος Γκέρχολτ. Παρακαλώ. Θα μας συνοψίσετε εσείς την πρόταση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που αντικαθιστάτε τον κύριο Μαρτουσέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, θα διαβάσω μία δήλωση του εισηγητή του κυρίου Μαρτουσέλο. Καταρχάς, ε, ζητεί συγγνώμη που δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει αυτοπροσώπως ε, τις ιδέες του και ευχαριστεί εμένα που τον εκπροσωπώ. Όσον αφορά το θέμα αυτό, τα μέτρα για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ε, ΦΠΑ είναι κάτι που συζητήσε εδώ, και, πολύ καιρό, διότι το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει και τα όρια του. Οι εργασίες μας θα ε, οδηγήσουν σε έναν καλύτερο και πιο απλό ε, κανονισμό. Το σύστημα που έχουμε εφαρμόζεται εδώ και αρκετέ ε, δεκαετίε ε, και δεδομένου των εξελίξεων στην κοινωνία και στην εσωτερική αγορά, οι ανάγκε είναι σαφεί. Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί με πολλού τρόπου και ανάλογα έχουν εξελιχθεί και οι προκλήσει. Ο εισηγητή λοιπόν πιστεύει ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανεί και Γι' αυτό είναι απαραίτητη μια καλή κατανόηση των προκλήσεων. Θέλουμε να διευκολύνουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και να μειώσουμε τις δαπάνες τους. Ο κύριος ε, Μαρτουσέλο χαίρεται που είναι εισηγητής για το θέμα αυτό και τονίζει ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές και το προσωπικό ε, θα οδηγήσει σε έναν καλύτερο κανονισμό που θα είναι πιο απλός, ε, διαφανής και θα συνδέεται με την αστερική αγορά που έχουμε δημιουργήσει. Όσον αφορά τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία, όπου βλέπουμε κάποιους περιορισμούς ε, σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τον αντίκτυπο. Και ο κύριος Μαρτουσέλο πιστεύει ότι πρέπει να περιορίσουμε την απάτη και να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της απάτης, να προστατεύσουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη από τον αρνητικό αυτόν αντίκτυπο. Προσβλέπει Μάλλον εγώ θέλω πολύ να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις όσον αφορά τις τροπολογίες και ο κύριος Μαρτουσέλο θα ξεκινήσει τις εργασίες του με βάση τις παρατηρήσεις σας. Ε, παραμένει στη διάθεσή σας ε, για οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων και σας ευχαριστεί που με ακούσατε. <laughs> Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ε, διαβάσατε την εισαγωγή του εισηγητή μας. Ο Γιέπε είναι η εισηγητής του S&D, είναι παρόν ο κύριος Τάγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Γέπε Κόφοθ ζητεί συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Θα μιλήσω λοιπόν εκ μέρους του. Η ομάδα S&D επικροτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ε, τις αναλυτικές προτάσεις όσον αφορά τους ακρογωνιαίους λήθους ε, για το μελλοντικό οριστικό σύστημα ΦΠΑ. Είναι σαφές ότι το ισχύον σύστημα είναι ανεπαρκές όσον αφορά την αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης. Ε, γι' αυτό επικροτούμε την πρωτοβουλία που στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις ε, αιτίες ε, και να περιορίσει τις ε, απάτες που ανέρχονται σε 41 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το ε, S&D θέλει αυστηρά κριτήρια που να εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να δούμε ποιες επιχειρήσεις μπορούν ε, να ε, λάβουν το καθεστώς ε, του πιστοποιημένου υπόχρεου ΦΠΑ. Η ομάδα S&D θέλει απόλυτη διαφάνεια και πιστεύουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερωθούν σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί το εν λόγω καθεστώς. Θα πρέπει να ασχοληθούμε περαιτέρω με τους φορολογούμενους ε, για να μην ε, έχουμε φοροαποφυγή. Επίσης, ε, ζητάμε από τον εισηγητή, σε συνεργασία με τους κοιόδες εισηγητές, να ξεκινήσουν επικοδομητικό διάλογο πάνω στις νέες μορφές απάτης που μπορεί να υπάρξουν αφού εφαρμοστεί το νέο σύστημα ΦΠΑ. Θέλουμε επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.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 Uh, Η συζήτηση λοιπόν θα γίνει ε, επί του σχεδίου εκθέσεως να σας πω δύο λόγια σχετικά με την έκθεση Ρωσάτη όσον αφορά την σημαντική ψηφιακή παρουσία. Υπάρχουν 110 ε, τροπολογίες στα 14 ε, του εισηγητού. Οι περισσότερες τροπολογίες ε, θέλουν να κάνουν την διασύνδεση με τις προηγούμενες προτάσεις CCCP καθώς επίσης και τις συμφωνίες περί φορολόγησης και τις αρχές του ΟΣΑ. Επίσης ε, ε, γίνεται λόγος ε, σε την ψηφιακή, σημαντική ψηφιακή ε, παρουσία καθώς επίσης και με την ρήτρα αναθεώρησης. 183 τώρα είναι οι τροπολογίες για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, τροπολογίες οι οποίες αφορούν κυρίως την, τα ψηφιακά interface σε την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, ε, την αύξηση ε, των ε, ποσοστών καθώς επίσης και την εισαγωγή μιας sunset, ρήτρας sunset. Ε, θα πρέπει να γίνει συμφωνία όσον αφορά τους, ε, τις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και αυτό μέχρι την 3η Δεκεμβρίου. Όσον αφορά το πρώτο θέμα για τις μακροπρόθεσμες λύσεις, ο κύριος Ροσάτη δυστυχώς δεν είναι εδώ, ίσως να έχει προσγειωθεί, ίσως να βρίσκεται ακόμα στους εθέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μιλήσει ο συνάδελφος εκ ονόματός του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα διαβάσω αυτά που μου έστειλε ε, ο κύριος Ροσάτη. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάγκα και τους κοιόδης συγητές για την εξαιρετική συνεργασία και την επικοδομητική, το επικοδομητικό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω επίσης την Γραμματεία για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει όσον αφορά το φάκελο αυτό. Στην ουσία ε, οι 120 τροπολογίες αλλά και οι 14 τροπολογίες του εισηγητού υποστηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά κατανοούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών ε, προτιμούν μακροχρόνιες ε, ε, λύσεις και θεωρούν το θέμα της φορολόγησης των εταιριών πολύ σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε τέτοιες μακροπρόθεσμες λύσεις ε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην εγκρίνουν μονομερείς λύσεις οι οποίες οδηγούν τέλος ε, σε κατακαιρματισμό της αγοράς καθώς επίσης και ε, ανασφάλεια. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την σημαντική τους συνεργασία. Στην προετοιμασία των συμβιβαστικών τροπολογιών ε, ε, προσπαθήσαμε να τις χωρίσουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Ε, στην πρώτη κατηγορία αυτές που δεν θέλουν την πρόταση της Κομισιόν και ο κύριος Ροζάτη της απορρίπτης. Δεύτερον, τροπολογίες οι οποίες κατά την άποψή τους δεν δίνουν μεγάλη δυνατότητα εξέβρεση συμβιβασμού με την πλειοψηφία. Κατηγορία 3, οι τροπολογίες επί των οποίων μπορούμε να στηριχτούμε για συμβιβασμό συμβαστικές τροπολογίες ε, και τέλος ε, οι, αυτές οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν ε, γιατί δεν αποτελούν προτεραιότητα στις πρώτες συναντήσεις των σκιοδών έγινε λόγος για όλα αυτά τα θέματα και ο εισηγητής χαίρεται γιατί μπορεί να πει ότι έχουν βρεθεί επί πολλών σημείων συμβιβασμοί. Υπάρχουν 11 συμβιβαστικές, ε, οι οποίες ενδεχομένως όμως να αλλάξουν ε, στην επόμενη συνεδρίαση. Οι 11 αυτές συμβιβαστικές ε, καλύπτουν ήδη την ε, κατάσταση που αφορά την, τριετή, ε, την πάροδο τριετούς ε, διαστήματος μέχρι την υποβολή έκθεσης. Επίσης υπάρχουν συμβιβαστικές οι οποίες αφορούν την, τα προσωπικά δεδομένα. Ο κύριος Ροζάτη βεβαίως θα είναι πάντα στη διάθεση των υπολείπων. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε τις δύο εκθέσεις μαζί. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω τον ε, λόγο ε, στον συνάδελφο που είναι ε, υπεύθυνο για τις πρόθεσμες λύσεις, ο οποίος όμως είναι και σκιώδης για τις μακροπρόθεσμες. Ευχαριστώ ε, πολύ. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Ρωσάτη σχετικά με τη φορολόγηση εταιριών με σημαντική ψηφιακή ε, παρουσία. Πρέπει να επιβεβαιώσω ότι η εργασία ε, έγινε σε πνεύμα συνεργασίας και βασιστήκαμε στην ενοποιημένη βάση και την κοινή ενοποιημένη βάση, CCTV, CCTV. Και έχουμε εκφράσει συγκεκριμένες ε, συστάσεις ε, οι οποίες αφορούν και το ευρωπαϊκό αλλά και τα εθνικά φορολογικά συστήματα. Επομένως, εμείς θέλουμε μια καλά δομημένη ε, προσέγγιση. Βεβαίως, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις όσον αφορά το πεδίο ε, εφαρμογής ε, και όσον αφορά το ευρύ πεδίο το οποίο θα περιλαμβάνει τις εταιρείε με σημαντική ψηφιακή παρουσία. Επίσης, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα των εταιρεών με σημαντική ψηφιακή παρουσία. Πάντω, η συνεργασία γίνεται ε, σε ε, καλό πνεύμα, πνεύμα συνεργασία και επομένω. Ε, για τα CCTB και τα CCTB η συζήτηση είναι πολύ, γίνεται σε πολύ καλό κρίμα. Επίση, ε, η συζήτηση δεν γίνεται μόνο για εταιρείε με σημαντική ψηφιακή ε, παρουσία, ε, αλλά και για τι για τις συγκεκριμένες ψηφιακές υπηρεσίες και επομένως εμείς εδώ θα θέλαμε κυρίως ε, να ε, αναφερθούμε στην ε, μη σωστή επιβολή φορολογίας σε γίγαντες της ψηφιακής σκηνής. Επ' αυτού βεβαίως σημαντική συζήτηση θα λάβει η χώρα την 4η Δεκεμβρίου. Ποια πρέπει να είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την παρούσα φάση. Ε, δεν έχουμε ακόμα συνάντηση για το DST με τους ε, σκιώδεις, ε, αλλά είναι γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση πρόσκαιρη. Οπωσδήποτε όμως και για το DST γίνεται συζήτηση και για το ψηφιακό περιεχόμενο. Έχουμε άλλες τροπολογίες οι οποίες αφορούν την πώληση online, επιγραμμική πώληση προϊόντων, αγαθών είναι 134, 135, 136 μέσω των οποίων διευρύνεται το ε, πεδίο εφαρμογής ε, ε, σημαντικά. Πραγματικά, αν το σκεφτεί κανείς σωστά, η παρούσα πρόταση της Κομισιόν μπορεί ας πούμε να εφαρμοστεί στο Facebook αλλά όχι σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της Amazon. Τέλος, ε, ε, συζήτηση για τα κατόφλια, πολύ σημαντική. Κάποια ε, μέλη πρότειναν τη διαγραφή αυτού του κατοφλίου των 50 εκατομμύριων ευρώ αλλά αυτό, το 50 συγγνώμη, αλλά αυτό έρχεται μαζί με κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να διαγραφούν. Εδώ γίνεται μια πρόταση μεταξύ των 25 και των 100 εκατομμυρίων να υπάρχει ένα ποσοστό 3% το οποίο θα αυξάνεται όταν περάσουμε τις 100.000. Ε, υπάρχει μία ε, τροπολογία, είναι η τροπολογία 158 και η τροπολογία 165. Εδώ ε, γίνεται μία προσπάθεια εισαγωγής ε, ε, κάποιων μέτρων προσωρινών. Πάντως το σημαντικό είναι να δούμε την κατάσταση και να προετοιμαστούμε ε, για περιπτώσεις όπου το βάρος μπορεί λόγω εσφαλμένων κινήσεων να αυξηθεί. Επανερχόμενο στη συζήτηση για την ρήτρα Sunset, μας μίλησαν και οι Υπουργοί για το θέμα αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, λέμε ότι αυτή είναι μια ε, πρόταση προσωρινή εν αναμονή πιο διορθωτικών λύσεων και επομένως κατά την έννοια αυτή θα μπορούσαμε να δεχτούμε ε, το SDP ή το CCTV γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει και το εθνικό σύστημα και το, και το ευρωπαϊκό σύστημα να προσαρμοστούν στην σημαντική ψηφιακή παρουσία. και οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτά τα προσωρινά μέτρα. Αυτά θα τα δούμε όμως στο μέλλον. Ε, βεβαίως το μέλλον είναι άμεσα, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα είδος DST ε, ήδη από τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από το ΕΛΚ, ε, είναι η εισηγητής ο Καπιέλ Μάτο για την έκθεση του Πολ Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μάτο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τις προτάσεις και τις εκθέσεις. Να, να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Μάτο που δεν μπορούσε να είναι εδώ, λέει η κυρία Λόπες Φοντανιέ. Ε, ε, είναι συντονιστής ε, του ΕΛΚ σε μια αποστολή αλίας κατά τον ε, κύριο Μάτο ο σχεδιασμός ενός σταθερού ε, φορολογικού πλαισίου είναι απαραίτητο έτσι ώστε ε, σε μια τόσο μεγάλη εσωτερική αγορά τόσων εκατομμυρίων καταναλωτών να υπάρξουν καλές βάσεις. Επίσης θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να, είναι, να δείξει ρεαλιστική στάση και να προσπαθήσει να βρει συνενετικές συμβιβαστικές ε, λύσεις. Ο καθένας θα πρέπει να πληρώσει αυτό που του αναλογεί, εκεί που του αναλογεί ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε επιγόντως να βρεθεί λύση έτσι ώστε ε, να πληρώσουν όλες οι επιχειρήσεις αυτούς τους φόρους που τους αναλογούν και να μην τα πληρώνουν πάντα οι παραδοσιακές ε, Επιχειρήσει Τέσσερα είναι τα κεντρικά σημεία. Ε, το πρώτο, ποιε είναι οι υπηρεσίε οι οποίε θα πρέπει να υπόκεινται σε αυτό το φόρο. Επίση, η πρόταση του 5% για την Κομισιόν. Τρίτον, ε, ρήτρα αναθεώρησης, πολύ σημαντικό θέμα. Και τέλος, τελευταίο σημείο, να διασφαλιστεί ότι αυτή θα είναι, αυτό θα είναι προσωρινό μέτρο και όταν θα βρούμε το τελικό μέτρο θα πρέπει να σταματήσει αυτή η φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Ο κύριος Μάτο δεν μπορεί να συμφωνήσει με την πρόταση του εισηγητού όσον αφορά το δεύτερο θέμα ε, που θέλει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογή ε, και να αυξήσει την φορολόγηση γιατί αυτά είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν και να αναλυθούν σωστά. Ορισμένες ε, χώρες μέλη όπως η Ισπανία ήδη ε, προχωρούν και προωθούν μια δική τους ε, πρόταση χωρίς όμως να διαβρύνουν το πεδίο εφαρμογής. Εάν αυξηθεί ε, το πεδίο εφαρμογής ή ο ίδιος ο φόρος θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδεχόμενο αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα θα είναι αναλογικά. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παίρνει τέτοιες αποφάσεις χωρίς να έχει τη βεβαιότητα των επιπτώσεων. Μια δυνατότητα θα ήταν να ζητήσουμε από την ε, Κομισιόν ε, μια αυστηρή ε, ρήτρα αναθεώρησης έτσι ώστε να δούμε εάν είναι βιώσιμα αυτά τα μέτρα ή αν θα είναι βιώσιμα τα μέτρα αυτά. Όσον αφορά το τέταρτο σημείο, ο κύριος Μάτο θεωρεί θεμελιώδου σημασία να συνεχίσει η καταβολή προσπαθειών έτσι ώστε ο ψηφιακός φόρος να είναι μονάχα και αποκλειστικά μεταβατικό μέτρο. Τέλος, ε, θέλει να υπογραμμιστεί η παρουσία και του Κοινοβουλίου στην διαδικασία αυτή ε, και η επικοδομητική συμμετοχή του σε αυτήν την συζήτηση. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το μέτρο θα ενισχύσει την ενιαία ψηφιακή μας αγορά και όχι να αποφασίσουν κάποιες χώρες μέλη να εφαρμόσουν δικά τους μέτρα ενώ άλλα κράτη-μέλη θα ε, εφαρμόσουν αυτήν την πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τους διαπραγματευτές για όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει. Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρου του ECR. Είναι σκιώδης η Ashley Fox, δεν είναι παρόν όμως. Από την άλλη έχουμε τον Πέτρι Γέσεκ, τον οποίο αντικαθιστά ο κύριος Τρεμόσα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ ως συντονιστής. Ε, θα πάρω το λόγο για τα δύο αυτά θέματα εκ μέρους του Πέτρι Γέσεκ που δεν έχει φτάσει ακόμα στις Βρυξέλλες. Όσον αφορά την έκθεση Ροζάτη, ε, σχετικά με την ε, σημαντική ψηφιακή παρουσία. Ε, επικροτούμε τη δουλειά που έχει γίνει από τον εισηγητή στο θέμα αυτό. Και συμφωνούμε με τις τροπολογίες που έχει υποβάλει ο εισηγητής. Ιδιαίτερα ο κύριος Γέζεκ χαίρεται που υπογραμμίζεται η σημασία του να σκεφτούμε προσεκτικά τα κριτήρια για να έχουμε την πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμη λύση. Ο σκιώδης μας επίσης ε, χαίρεται που ε, βλέπει να σεβόμαστε την ακαιρεότητα των ε, μικρών επιχειρήσεων. Επικροτεί την πρόταση των ε, συναδέρφων ε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει αν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες σε τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ ε, της οδηγίας. Προσλέπει στην περαιτέρω συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά και είναι πεπισμένος ότι σύντομα θα βρεθεί συμβιβασμός. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, όπου η συγκητής είναι ο Πολ Τάγκ, θα σας διαβάσω τις παρατηρήσεις που μου έστειλε πριν λίγα λεπτά. Όπως ε, ήδη είπε ο Πίτρη Γιάζεκ σε προηγούμενες συζητήσεις, επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην έκθεση αυτή, καθώς και τις τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής ε, και οι σκιώδεις εισηγητές στο θέμα αυτό. Ιδιαίτερα, επικροτεί τα εξής ε, στοιχεία. Καταρχάς, το να διασφαλιστεί τα κριτήρια να είναι επαρκή, ώστε καμία επιχείρηση ε, να μην πέσει στο κενό. Και γι' αυτό επικροτεί την πρόταση των άλλων σχεδόν εισηγητών ε, να γίνει αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο χρόνια μετά την ε, έναρξη ισχύω της οδηγίας αντί για τρία χρόνια. αυτό έχει να κάνει με το άρθρο 24 και τον σχετικό συμβασμό. Ο Πίτερ Γιέζεκ επίσης επικροτεί το ότι ο εισηγητής συμμερίζεται τη θέση ότι η φορολογία θα πρέπει να περιορίζεται σε επιχειρήσεις με συνολικό τζίρο σε όλο τον κόσμο 750 εκατομμύρια ευρώ, διότι έτσι περιορίζεται ο αντίκτυπος ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, κάποιοι συνάδελφοι ε, θέλουν να ε, συμπεριλαμβάνονται εδώ οι επιχειρήσεις ε, με ε, έσοδα στην Ένωση άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμω μπορεί να είναι προβληματικό για, κάποιες, για κάποια κρατημέλη, διότι θα είναι ιδιαίτερα επαχθή ο ορισμός αυτός. Γι' αυτό προτείνεται μια ενδιάμεση λύση, μια προσωρινή λύση. Ο Πίτερ Γέζεκ συμφωνεί η σημαντική ψηφιακή παρουσία να περιοριστεί στι επιχειρήσεις ε, με κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ε, συμφωνεί σε μια τροπολογία που πρόσφατα υποβλήθηκε από συναδέρφους την πρόταση για το 5% της φορολογίας ε, για έσοδα άνω των 100 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Ιέζεκ πιστεύει ότι κάποιες, ε, κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο δεν μπορούν να δεχτούν την πρόταση αυτή. Κάτι όμως που, δεν μπορούμε να, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, διότι θέλουμε να καταλήξουμε συμβασμό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Προτείνεται λοιπόν ο φορολογικός συντελεστής να είναι 3%. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόζα που μας παρουσιάσατε τις θέσεις ε, του Πέτρι Γιέζεκ. Η Εύα Ζόλη που είναι η συγκήτρια του Πρασίνων δεν είναι παρούσα. Η κυρία Σκοτ Κέιτο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα καλύψω και τις δύο εκθέσεις για την έκθεση του κυρίου Ροζάτη. Συναδελφός θέλω να τον ευχαριστήσει για το μέχρι τώρα έργα του και να τονίσει δύο-τρία στοιχεία. Η ομάδα μας καταρχάς θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό άπαξ και δοθεί ένα συγκεκριμένο ορισμό τη ψηφιακή παρουσίας να ενσωματωθεί σε όλες τις διμερείς ε, συνθήκες για φορολογικά θέματα για να μην μείνουν παραθυράκια και γι' αυτό ζητούμε από το Συμβούλιο τη σχετική τροποποίηση της εντολής τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναδιαπραγμάτευση φορολογικών συμφωνιών με τρίτε χώρε για να έχουμε ένα πλήρε ε, φορολογικό περιβάλλον. Παρακαλώ και του λοιπού και να εξετάσουν ε, το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν την πρόταση αυτή. Ε, για την βραχυπρόθεσμη εφαρμογή της οδηγίας τώρα για, τους, για την φορολογία θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να αρκέσει μια προσωρινή εφαρμογή για να καλύψει τα προβλήματα στη φορολογία των ψηφιακών επιχειρήσεων. Τρίτον, ε, γνωρίζοντα βέβαια ότι υπάρχει πολιτική διαφωνία, θέλουμε να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο φορολόγηση, ένα ελάχιστο συντελεστή φορολόγηση, χωρίς το οποίο θα εξακολουθήσουν τα προβλήματα σχέση με τον ε, φόρο επιχειρήσεων και μπορεί και να επιδεινωθούν. Αυτές είναι οι σκέψεις μας σε σχέση με τα θέματα του κύριου Ροζάτη για τον κύριο Τάγκ, ευχαριστώ τον και πάλι για τη δουλειά του μέχρι τώρα. Ή υποστηρίζουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να καλύψει πλατφόρμες όπως το Netflix και το Amazon και ε, με το σκεπτικό ότι σε ένα ψηφιακό κόσμο είναι πολύ δύσκολο να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ του χρήστη και του ε, πελάτη, γιατί και οι δύο μπορούν να συμβάλλουν στην προσθεμένη αξία μιας ψηφιακή επιχείρησης. Υποστηρίζουμε την αύξηση του DST από το 3% στο 5%. Συμφωνούμε με τον εισηγητή δηλαδή ότι το περιθώριο που είχε προβλεφθεί για τις ψηφιακές επιχείρησεις ήταν πολύ περιορισμένο, πολύ μετριοπαθές από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ε, συμφωνούμε με όλους τους σκιώδες εισηγητέ ε, σε σχέση με τα 275 εκατομμύρια ευρώ που θέλουμε να, διακρι... να διαγράψουμε. Τα 15 πρέπει να παραμείνουν έσοδα από τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το δεύτερο κατόφλι είναι το σημαντικό πιστεύουμε για το θέμα αυτό και μπορεί να επιτρέψει την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από υπερβολικές απαιτήσει. Τελευταίο και σημαντικό στοιχείο είναι να ασκηθεί πίεση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε μια μακροπρόθεσμη λύση να ε, εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό και να εφαρμοστεί για να επιτευχθεί το δυνατόν ε, ευχερέστερα μια συμφωνία πρέπει να επικαλωστούμε το άρθρο 116 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διαδικασία της συναπόφασης και την ειδική πλειοψηφία. Ξέρουμε βεβαίως ότι ο Γιουνκέρι, ο Μοσκοβισή ως μέλος Επιτροπής έχει υποσχεθεί ότι θα αντιμετωπίσει υπό το 116 φορολογικούς παραδείσους και πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή να τηρήσει την υπόσχεσή του αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη ε, συμφωνία για τα δύο αυτά θέματα και να αποδείξουμε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει αποτελέσματα εγκαίρω για τα θέματα των φορολογικών παραδείσων, αντίθετα από τα κράτη-μέλη που παρεμποδίζουν ακόμη τι επίδοση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλοι από την ΚΟΕ, του. Ε, DD και του CNF δεν έχουμε σκιώδεις ηγητές. Θέλει κανείς να λάβει το λόγο σε διαδικασία καρστία ή όχι. Ο Πολ Τάγκ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, πολύ σύντομα. Για να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ή εκπροσώπους αυτών για τα σχόλιά τους. Για τον Διεστή. αυτό πρέπει να κοιτάξουμε είναι να μην ε, ξεκινήσει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της χωριστά ε, το Ρωμανό Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να διαφυλαχθεί η ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς η οποία ταυτόχρονα απαιτεί να συζητηθεί τόσο το πεδίο όσο και ο συντελεστής γιατί έτσι έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Οπωσδήποτε χρειάζεται αυτό. Και άρα πρέπει να συστήσουμε και το πεδίο εφαρμογή και το συντελεστή. Και μετά το θέμα είναι ότι αν ζητούμε αξιολόγηση επιπτώσεων, αυτό θα αποδειχθεί δύσκολο καθώς είμαστε σε χαρτογράφητα νερά. Θα χρειαστεί πολύ πολιτική βούληση και βεβαίως χρειάζεται μια ταχύτατη επισκόπηση αλλά αξιολόγηση συνεπειών ίσως δεν είναι η κατάλληλη λύση. Αυτό που κάνουμε λοιπόν όταν πιέζουμε το TST και όλα τα λένε ότι καταφέρουμε να φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ΗΠΑ. Στο BEPS πρώτο πρόγραμμα και πρώτη δράση ήταν η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Ανεβλήθη όμως, άρα πρέπει το Κοινοβούλιο να πιέσει για μια όχι μόνο ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή λύση στο θέμα αυτό. Τέλος συμφωνώ πως χρειάζεται πλέον η Ευρώπη να πραγματοποιήσει πρόοδους όχι μόνο για το DST αλλά και για το CCTV και για όλα τα άλλα ζητήματα και χρειάζεται ε, ειδική πλειοψηφία διαδικασία συναπόφασης οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μεγαλύτερες σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε τις εξουσίες επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνατότητα δράση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με πλειοψηφική απόφαση και όχι με ομοφωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμασού. Πρόεδρε, ευχαριστώ να μου επιτρέπετε να λάβω το λόγο μετά τον εισηγητή στα αγγλικά αλλά στα γαλλικά τώρα θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε ο Πολ το εγχείρημα για την ψηφιακή οικονομία, του DST, πρέπει να προλάβουμε την εξέλιξη κατά την οποία ορισμένες χώρες ε, εισάγουν δικά τους συστήματα φορολογίας που θα, θα γελιοποιηθούν, θα αποτύχουν σε τελευταία ανάλυση, θα είναι πολύ περιορισμένα φορολογικά συστήματα και σε όγκο. Και όπως είπε ο Πολ, μας ενδιαφέρει και το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, να έχουμε το ίδιο φορολογικό σύστημα στον τομέα αυτών για όλους, νέο φορολογικό σύστημα, νέα τεχνολογία σε τελευταία ανάλυση. για την ε, εσωτερική αγορά. Και όπως είπε και ο Πολτάγκ, θα προσθέσω και εγώ, ότι στις μελέτες επιπτώσεων που βεβαίως θα χρειαστούμε, αλλά δεν θα μπορούμε να τις εξασφαλίσουμε γιατί ούτε στο Συμβούλιο δεν καταθέτουν τις ε, τα πορίσματά τους στα κράτη-μέλη. Προφανώς αυτό είναι πολύ δυσάρεστο, μας φέρνει στη δύσκολη θέση να πρέπει να κάνουμε προτάσεις χωρίς να ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει. Πληροφορίες σε σχέση με την απόδοση σε όγκο περιορισμένο δισεκατομμυρίων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία μάλλον θα έχει να κάνει με 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ απόδοση φορολογική το χρόνο, δηλαδή οικονομικές συνέπειες όχι τεράστιες. Ούτε τραγικέ ούτε και ως προ το θετικό των, ε, των εσόδων που μπορεί να φέρουν. Τώρα για τη μακροπρόθεσμη πρόταση και την ε, έκθεση Ροζάτη το να θέλουμε όσα να γνωματεύσει πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε απλώς παρέλκυση για αυτούς δηλαδή που δεν θέλουν την εισαγωγή φορολογίας. Σημειώνω δε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μόλις πριν από ένα χρόνο εισήγαγαν Μίζωνα φορολογική μεταρρύθμιση που αφορούσε και τον άμεσο φόρο, που αφορά του ιδιώτε και αυτό δεν είναι σχετικό με το δικό μα θέμα, αλλά και το φόρο των επιχειρήσεων που έχει άμεση συνάφεια με αυτά που συζητούμε, χωρί να συζητήσουν που δίνει το ενδεχόμενο να τους ενδιαφέρει στο πλαίσιο του ΟΣΑ να συζητήσουν μαζί μας ή με άλλους το πώς θα διαμορφωθεί το αμερικανικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, αν το θέλουμε και οφείλουμε νομίζω να το πράξουμε, να συζητήσουμε στο πλαίσιο του ΩΣΑ με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και άλλους, γιατί δεν είναι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείες, πρέπει εμείς πρώτα να έχουμε εισαγάγει το δικό μας σύστημα, το ευρωπαϊκό σύστημα, τις δικές μας θέσεις και από εκεί και πέρα μπορούμε ισότιμα να συνομιλήσουμε ιδάλλως ή δεν θα εισαγάγουμε σύστημα δικό μας ή θα είμαστε καταδικασμένοι να ακολουθήσουμε αυτό που έχουν ε, εισαγάγει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ πολύ, Άλαν. Άλεν. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι θα πρέπει ε, οπωσδήποτε όλη η Ένωση να προχωρήσει ε, σε αυτήν την ε, πρόταση. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν θα είναι σωστό είτε από άποψη φορολογική είτε από άποψη ισοτιμίας της αγοράς κλπ. Το Κοινοβούλιο είναι σαφέ ότι μέσω εισηγητών και σκιωδών ε, θα προωθήσει τη θέση του προ το ε, Συμβούλιο. Έχουμε τώρα ε, ένα επόμενο σημείο, αλλά φοβούμε ότι θα πρέπει πάλι να διακόψουμε για 10 λεπτά ή και λίγο περισσότερο, έτσι ώστε να έρθει και η εισηγήτρια του επομένου σημείου. 16 λοιπόν και 15 θα είμαστε ε, εδώ ε, ξανά έτσι ώστε να μελετήσουμε την έκθεση της κυρίας ε, Σάντερ όσον αφορά την πρόθεση της χρήσης αγορών ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα. Ε, έχουμε 20 ε, λεπτά ε, για την πρόθεση της χρήσης αγορών ανάπτυξη σε ΜΜΕ. Η συγγήτρια είναι η Αν Σάντερ από το ΕΛΚΑ και μιλάμε για την εξέταση των τροπολογιών, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, η οποία καλύτερα από μένα μπορεί να εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σκιώδης εισηγητέ για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και να τις ευχαριστήσω επίσης και για την καλή συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων που μέχρι τώρα έχουμε κάνει. Το κείμενο αφορά ε, ε την ε, πρόθεση της χρήσης αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ε, μπορεί να αποτελέσει την δυνατότητα πρόθεσης των πλατφορμών ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα τρεις πλατφόρμες έχουν δημιουργηθεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν, αν θέλουμε να εθαρρύνουμε την κίνηση αυτή, να προβλέψουμε επιπλέον ελαφρύνσεις έτσι ώστε να προσελκύσουμε περισσότερες μικρομεσαίες σε αυτήν την αγορά αλλά και για να δώσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξη νέων πλατφορμών. Όπω επανειλημμένα έχω πει, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% των ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη και παίζουν και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση τη ευρωπαϊκή οικονομία μετά την κρίση. Υπάρχουν προγράμματα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αλλά συχνά βλέπουμε ότι δεν, λαμβάνουμε, δεν λαμβάνονται επαρκώ υπόψη οι ιδιαιτερότητε αυτών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ιδίω δε όσον αφορά το χρηματοδοτικό κομμάτι, όπου λίγε ελαφρύνσει προτείνονται διότι υπάρχει πάντα κίνδυνος κατακαιρματισμού. Εάν ε, θέλουμε να κατανοήσουμε αυτήν την... Ε, μπορούμε να κατανοήσουμε βέβαια αυτήν την ε, ανησυχία, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο περισσότερο ελαφρύνσεως, πράγμα που προβλέπεται στο κείμενο. Έχουμε προχωρήσει ήδη. Έχουμε κάνει δύο συνεδριάσεις με τους κοιόδης συγητές μία τεχνικής φύσεως σήμερα το απόγευμα και ίσως να σας πω ε, δύο λόγια όσον αφορά το πόσο έχουμε προχωρήσει, όσον αφορά τις συζητήσεις μας. Νομίζω ότι προχωρήσαμε καλά επί αρκετών ε, σημείων, όπως ας πούμε ε, τα, οι, οι συμβάσεις ρευστότητας ή οι ρήτρες αναθεώρηση που αφορούν διάφορες τομεακές νομοθετήσεις. Ναι, θελήσαμε να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα ε, σε σημεία στα οποία υπήρχαν φαιές ζώνες όσον αφορά την νομοθεσία. Σήμερα παραμένει ένα ερώτημα, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, ζήτημα το οποίο αφορά τους ε, καταλόγους ε, που θα πρέπει, οι που θα πρέπει να δοθούν εις τις αρχές, καθώς επίσης και ε, την αιτιολόγηση μεταφοράς ε, της ε, πληροφόρησης. Υπάρχει μια άποψη η οποία λέει ότι αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις στέλνει ε, η ε, επιχείρηση και θα πρέπει να είναι σε θέση να τις ε, δίνει στην αρμόδια εθνική αρχή εάν αυτή η αρχή τη ζητήσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη που λέει ότι αυτές οι πληροφορίες, θα, οι προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να στέλνονται έτσι κι αλλιώς. Εγώ ε, λέω ότι περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται μονάχα μετά από συγκεκριμένο αίτημα, διότι εάν συστηματικά ε, στέλνονται στην αρμόδια αρχή οι πληροφορίες, τότε θα αναγκαστούμε ε, να ε, έχουμε πιο αυστηρές ε, διαδικασίες και προϋποθέσεις σε αυτές τις αγορές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι στις κεφαλιακές αγορές. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ξαναδούμε. Ίσως υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο που αφορά ε, τα κατόφλια χωρίς όμως ε, να αγγίξουμε το μύφι ή το γιατί είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα τελικές θέσεις. Ε, αυτά συζητήσαμε με τους δύο δεσίγητες, ε, τους οποίους θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω σήμερα εδώ ενώπιόν σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας αυτή, καθώς και τις πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Η Νίνα Γκίλη Νεσκιώδης από το S&D, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Αν για την έκθεσή της και την παρουσίασή της, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό βήμα το να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις κεφαλαίες αγορές και είναι κάτι που ζητάει η πολιτική μου εταιρεία, η πολιτική μου ε, ομάδα ήδη από την εποχή του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο του, ε, της οδηγίας ε, προσπέκτους. Είχαμε κάποιες ε, συνεδριάσεις της, ε, συναντήσεις της ομάδας εργασίας για το θέμα αυτό και είμαι ευγνώμων που γενικά έχουν ληφθεί υπόψη οι τροπολογίες μου στις συμβαστικές προτάσεις ε, της εισηγήτριας. Στόχος των τροπολογιών μου, κύριε Πρόεδρε, ήταν να διασφαλίσω την ισορροπία ανάμεσα στην καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τη και την προστασία των επενδυτών από την άλλη. Και στις συμβαστικές προτάσεις νομίζω ότι έχουμε σχεδόν βρει την σωστή ισορροπία. Επίσης, συμφωνώ με την μείωση του περιτού γραφειοκρατικού άχθους. Από την άλλη όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό οι εθνικές αρμόδιες αρχές να ενημερώνονται ψηφιακά. Το πιο επίμαχο για μένα θέμα, μάλλον, είναι ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενώ εκτιμώ την ανάγκη για αύξηση του κατοφλίου σε σχέση με τον, την ισχύουσα οδηγία MIFID, ε, με απασχολεί πολύ το να προχωρήσουμε από τα 200 εκατομμύρια στα 750 στο σημείο αυτό νομίζω ότι η ομάδα μου θα ζητούσε μεγαλύτερη επιφύλαξη. Διότι αλλάζουμε τους ορισμούς χωρίς να σκεφτούμε τις συνέπειες. Ναι, θέλω να δώσω περισσότερα κίνητρα, ωστόσο γίνεται περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Ωστόσο, σε κάποια κράτη-μέλη, εάν ανέβουμε στα 750 εκατομμύρια, τότε μιλάμε για τον ε, μεγάλο όγκο των ε, επιχειρήσεων στις χώρες αυτές, ε, οπότε ουσιαστικά στρεβλώνουμε τον, τον ε, ανταγωνισμό. Κάτι τέτοιο λοιπόν μπορεί να υπονομεύσει τις εργασίες που έχουμε κάνει σχετικά με την φόρο αποφυγή, διότι έτσι θα δημιουργήσουμε παραθυράκια στην νομοθεσία. Και μπορεί έτσι να δημιουργήσουμε και σύγχυση σχετικά με την επιλεξιμότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης. Εάν ε, λοιπόν τροποποιήσουμε τα κατόφλια θα πρέπει να φροντίσουμε να περιορίζονται στον τομέα αυτών και αυτό να μην γίνει εις βάρος της χρηματοδότησης των μικρότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτός ε, λοιπόν είναι ο βασικός ε, συμβασμός που θα πρέπει να πετύχουμε στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στην ολοκλήρωση των εργασιών. Νίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε κανέναν παρόντα από το ECR. Έχουμε όμως τον κύριο Τρεμόζα από την Άλτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σαντέχ για τη δουλειά της και το πνεύμα συνεργασίας με όλους τους ε, σκιώδες της. Έχει σωστά αγγλικά, διότι δεν είναι τόσο καλά τα γαλλικά μου, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλοί από εμά προέρχονται από διάφορες ε, περιφέρειες με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ εκπρόσωπω την ε, Καταλωνία με 8.000 πολυεθνικές, αλλά 500.000 μικρομεσαίες. Και όπως είδατε και σε άλλα σημεία της Ένωσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επομένω, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά Νίνα και την Επιτροπή, την και την Επιτροπή γιατί εξασφαλίζεται έτσι πρόσβαση στην κεφαλαϊκή αγορά για τι μικρομεσαίες. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης Πώ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ε, το ίδιο επίπεδο ε, τις ίδιες δυνατότητες ανάλογα με τη χώρα στην οποία εδρεύουν ε, στη χρηματοδότηση μπορεί να έχουν πρόσβαση στις ε, βόρειες χώρες της Ευρώπης πολύ ευχερέστεροι οι μικρομεσαίες από ότι στη νότια επί όπου μπορεί να έχουν μόνο μία πηγή χρηματοδότησης δηλαδή τον τραπεζικό δανεισμό γι' αυτό έχει σημασία να προχωρήσουμε σε εναρμόνιση αλλά και σε διάδοση και επέκταση των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ένωση. Οι επιμέρους συμβαστικές ε, τροπολογίες λοιπόν στην υπαριθμόν 1 ζητούμε ενίσχυση του ρόλου της ΕΣΜΑ που πιστεύουμε μπορεί να συμβάλλει με την πραγματογνωμοσύνη της ε, σημαντικά. Ως φιλελεύθεροι συμφωνούμε με όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, υποστηρίζουμε την συγγήτρια. Στη Β όμως θα θέλαμε και να το δούμε στην αυριανή μας συνεδρίαση ε, θα προτιμούσαμε να μείνει το πρώτο κείμενο, το πρώτο σχέδιο κειμένου, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο. Στη ΔΕΣΥ, όπως είπε και η Νίνα, δεν θέλουμε να φέρουμε επιπλέον ε, γραφειοκρατία ή επιβάρυνση γενικά για τις μικρομεσαίες με την εισαγωγή αυτών των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων που θα τις επιβαρύνουν για να έχουν ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ας το διευκρινίσουμε αυτό και με την τροπολογία C, τη συμβαστική. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι. Στην ε, παραδείγματι, έχουμε το θέμα των ε, της έκδοσης ομολογιών για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ε, ε, ρευστότητα, να μπορούν να μπουν δηλαδή στην αγορά της ανάπτυξης. Ας τα δούμε αυτά όλα αύριο. Ελπίζω ότι θα έχουμε πλειοψηφίες και συνένεση γενικά για να ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρομέουσα. Πράσινο σκιώδη δεν έχουμε. Η κυρία Λόπες όμως της Γκουέ είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαντέρα για την εργασία της και για την προσπάθεια ε, να ενσωματώσει και άλλες απόψεις ε, σε αυτό το τόσο τεχνικό θέμα. Ε, το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται πολύ και νομίζω ότι με τις τεχνικές προσαρμογές δεν θα βελτιωθεί. Θα χρειαζόταν μια πραγματική αλλαγή στην ίδια την αντίληψη του προγράμματος. Κατά την έννοια αυτή, εδώ δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε και πολλές προσδοκίες. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των ΜΜΕ όσον αφορά το μηχανισμό χρηματοδότησης, γιατί αποτελούν σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά την διατήρηση της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την πληροφόρηση, είναι αυτό και την επικοινωνία είναι σημαντικά θέματα. Επίσης θα πρέπει να ενδυναμωθούν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι εγγυώνται ότι δεν θα τεθεί ε, σε κίνδυνο η ιδιοκτησία όταν προσφεύγει κανείς σε τέτοιε μορφές χρηματοδότηση. Από την άλλη πλευρά πιστεύουμε ότι ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτές και να μην αφήνει καμία αμφιβολία σχετικά με ποιε είναι και ποιοι είναι ε, αυτοί και ποιοι είναι οι τρόποι με, τον, με τους οποίους μπορεί να προσφύγουν σε αυτήν την ε, χρηματοδότηση γιατί διαφορετικά ε, μπορούν να δημιουργηθούν, να προκληθούν οι κίνδυνοι που μπορούν να σχετίζονται ενδεχομένως και με την έλλειψη διαφάνειας σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσει διοικητικέ τέλο. ο ρόλος του εθνικού ρυθμιστή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είναι ε, διαφανής και ε, ε, δημόσιος, καθώς επίσης να μην δημιουργεί πρόβλημα και να θέτει ένα αμφιβόλο το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά, αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να βελτιωθεί το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω εάν ε, η εισηγήτρια θέλει τώρα να πάρει το λόγο. Όχι, δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους συναδέλφους και αύριο θα τα πούμε έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας όσον αφορά ε, τα θέματα ε, που μας απασχολούν. Επίσης και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ και αξιολογώ πολύ θετικά ε, την ε, κατάσταση. 3 ε, Δεκεμβρίου συζήτησε την Επιτροπή, στην Ολομέλεια δεν ξέρουμε πότε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το σημείο υπαριθμών 7 και χωρίς καμία διακοπή μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή το καθορισμό του προγράμματος Φισκάλης για την συνεργασία στον τομέα της φορολόγησης. Η συγητής μας ε, είναι ο Σβέν ε, Γκίγκολτ. Έχουμε πολλέ τροπολογίε 77 από άλλου υπόλοιπε από, 77 από άλλους ε, συναδέλφου, οι υπόλοιπε από τον ίδιο τον εισηγητή. Όμως καλύτερα να δώσω το λόγο στον εισηγητή και μετά θα ακολουθήσουν οι σκιώδει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο να σας ενημερώσω ότι έχουν διανεμηθεί οι συμβαστικές τροπολογίες. Έχουμε προχωρήσει καλά ε, και ικανοποιητικά. Πολιτικά νομίζω είναι πολύ βαρετή η έκθεση σε αντίθεση με τη σημασία του ζητήματος. Εδώ λοιπόν και όπως επιβάλλουν οι καλές παραδόσεις στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να βοηθήσουμε την καταπολέμηση της φοροαπάτης, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και στο πνεύμα αυτό διτυπώνονται και οι τροπολογίες. Χαίρομαι που βλέπω σε όλο το πολιτικό φάσμα πριν μια εξαίρεση που θα αναφέρω αργότερα ότι γίνονται δεκτές οι κύριες ε, ιδέες της έκθεσης φυσκάλης. Έχουμε συνομιλήσει και με τους εμπλεκόμενους ε, παράγοντες με κάποιες μικρές τροποποίησεις από πλευράς τους. Εν γέννη πάντως οι ιδέες έχουν ε, υποστηριχθεί και έχω λάβει υπόψη όλες τις προτάσεις των συναδέλφων. Ιδιαίτερα ζητήματα λοιπόν η διαφωνίες δεν είχαμε προς την ενίσχυση της ε, διαφάνειας του ε, ε, κειμένου και επίσης η αναφορά στις ειδικέ επιτροπές. Λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει αυτή η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών και σύγκληση έχουμε και στην ιδέα ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τον προπολογισμό προσαρμόζοντας τις προτάσεις της δημοσιονομικής με το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο γενικώ. Η ECR, αλλά δυστυχώ δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι, γιατί θα έξω το να το συζητήσουμε, δεν υποστήριξε ως ομάδα την πρόταση για υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να συμβάλλουν και αυτές σε πολυμερή συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων. Θλιβερό, γιατί ήδη υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα στο οποίο δυσκολεύονται να ενταχθούν ορισμένες από τις αναμεινωμένες χώρες και ενώ έχουν τη σχετική τεχνογνωσία τα ευρωπαϊκά κράτη και μπορούν να τις βοηθήσουν και πέραν ε, του ε, του 27-28. Βλέπω όμως ότι το ECR δεν, δεν υποστηρίζει την πρόταση αυτή. Θα ήταν καλό όμως ε, να μπορέσουμε να ε, συμβάλλουμε και στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων στο πρόγραμμα Φισκάλης. Δυστυχώς εκείνοι που έκαναν που διατύπωσαν τα πιο θεμελιώδη ερωτηματικά στο, για το πρόγραμμα αυτό δεν είναι εδώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα έχουμε συνεδρία των σκιωδών στις 20 Νοεμβρίου, ε, αφού βλέπω να επικρατεί γενικά υποστήριξη, το αφήνουμε σε επίπεδο τεχνικό, σε επίπεδο προσωπικού και αν δεν υπάρχει διαφωνία ψηφίσουμε στις 27 Νοεμβρίου για να πάμε στην Ολομέλεια αφού είναι κομμάτι του πολιτής δημοσιονομικού πακέτου και χαίρομαι γιατί έτσι όπως και άλλες επιτροπές που έχουν θέματα του πολιτισμού νομικού πλαισίου και εμείς ε, θέτουμε ψηλά τον πύχη για την ε, ταχύ επεξεργασία των ζητημάτων του μας. Το Φισκάλις έχει αποδείξει την ε, καλή του προσθέμενη, την υψηλή του προσθέμενη αξία και νομίζω μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς στη βελτίωση της έτσι περαιτέρω. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και εγώ που μας παρουσιάσατε μια καλή έστω και ε, βαρετή έκθεση. Ο κύριος Στόιαν δεν είναι εδώ. Παρακαλώ, ο κύριος Λαμασούρ. Ναι, αλλά θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση αν ήξερα την θέση του συναδέλφου Στρογιάν. Εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι συμφωνώ με την φιλοσοφική τοποθέτηση ε, του συναδέλφου και σίγουρα αστιεύεται όταν λέει ότι το θέμα αυτό είναι βαρετό, διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο από πολιτικής απόψεω και φυσικά από οικονομική είναι ε, θεμελιώδου σημασία, είναι ε, μίζωνος σημασία και πρέπει να το προωθήσουμε. Η η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, ε, φορολογικών ε, μηχανισμών κλπ. είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα ε, και η ευρωπαϊκή διαδικασία προς το πρέπει να ολοκληρωθεί σε αυτήν την θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου παρότι δεν ήταν προγραμματισμένη. Έχουμε τον κύριο Μπαγιέ από το S&D. Παρακαλώ. Ε, ναι, εγώ όμως είμαι συντονίστρια και επομένως εγώ θα κάνω τον σκιώδη του σκιώδους, λέει η κυρία περβάνς Μπερέσα. Θα δούμε πώς ε, ε, διαφαίνονται οι, και διατυπώνονται οι συμβιβαστικές. Ένα σημείο ε, το οποίο μας ενδιαφέρει είναι εάν οι δικές μας απόψεις έχουν ε, ενταχθεί, ενταχθεί συγγνώμη, σωστά. Αυτό που είναι σημαντικό για μας ε, βέβαια είναι η διάθεση με τα, στοιχεία 4, 5, 6 καθώς επίσης και το θέμα της φορολογίας των επιχειρήσεων όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων, την πληροφόρηση των διοικητών, λογισμικό κλπ. Τρίτη προτεραιότητα είναι η δυνατότητα, η προσπάθεια υπέρβασης των δυσκολιών ε, στην εφαρμογή του φυσκάλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, βεβαίως μας ενδιαφέρει ε, ένα είδος αντιπροσώπευσης των φορολογικών διοικήσεων στις Βρυξόλες, έτσι ώστε να σπάσει ο πάγος κατά κάποιο τρόπο των διοικήσεων που λόγω ε, ε φύσης αλλά και τάσης δουλεύουν σε κλειστό θάλαμο. Είναι πολιτισμική η διαφορά δηλαδή. Επίσης, το 74, το τροπολογείο 74, επιμένουμε σε αυτήν ε, και επιμένουμε και στο αντίστοιχο εκτιμώντας, διότι ε, στα πλαίσια αυτού, του σεμιναρίου ε, των διαφορείων, όπου θα συναντώνται οι διάφορες ε, διοικήσεις, θα πρέπει να έχουμε και εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων ε, γιατί έχουμε κατανοήσει ότι ε, γνωρίζουν τα συνδικαλιστικά όργανα και τα διακυβεύματα αλλά και τους κινδύνους. Ε, επομένως η άποψή τους και η συνεργασία με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων μπορεί να είναι θετική. Επίσης, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, στα πλαίσια της ανεξαρτησίας πάντα και επαφές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με εμά έτσι ώστε να γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τη συνεργασία. Βεβαίως μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, το είπαμε αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε με τον εισηγητή και επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ψηφιοποίηση, η διαδικασία ψηφιοποίησης και η πρόοδος της ε, ψηφιακής οικονομίας παραμένει πρόκληση που δεν θα ε, λυθεί μέσα από ένα απλό πρόγραμμα φυσκάλης. Οπωσδήποτε όμως ε, το φυσκάλης θα πρέπει να προσαρμόσει τα εργαλεία του σε αυτήν την ψηφιοποίηση της οικονομίας και επομένως να αντιμετωπίσει αναλόγως και τις δυνατότητες φορολογικής απάτησης. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε ε, εισηγητή του ECR που είναι πολύ κρίμα όπως είπε ο κύριος Γκίκολτ. Έχουμε όμως τον κύριο Τρεμόζα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ως συντονιστής ε, θα είμαι ο σκιώδης του σκιώδους. Ε, σκιώδης μας είναι η Καρολίνη Ναχτεχάου. Και θα μιλήσω γερμανικά. Η Καρολίνε μου είπε ότι έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά. Σε συγχαίρω λοιπόν. Και θα σας διαβάσω τις παρατηρήσεις που μου έδωσε. Είναι πολύ καλή και θετική η έκθεση αυτή. Έξι στόχους έχουν οι φιλελεύθεροι στις τροπολογίες που έχουμε προτείνει. Καταρχάς, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που συνδέονται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, θα πρέπει να αναλυθούν και δράσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η δεύτερη παρατήρηση της Καρολίνε είναι ότι τα μέτρα κατά της απάτης που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη ατομικά μπορεί απλά να μεταφέρουν το πρόβλημα σε γειτονικές χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει τις δράσεις. Τρίτον, ε, τα δημοσιονομικά θέματα θα πρέπει να επιτρέψουν εξυγχρονισμό των εργαλείων για την ε, υποβολή εκθέσεων ε, ώστε να εφαρμοστούν με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι φιλελεύθεροι είναι υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού σε 338 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια αύξηση ζητήσαμε στην ενδιάμεση έκθεση που υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης θέλουμε να αυξήσουμε τον ε, κατάλογο των επιλέξιμων δράσεων και τέλος δεν θέλουμε να ε, έχουμε πολλές εκθέσεις, να έχουμε μια ενιαία αιτήσια έκθεση ε, από κάθε κράτος μέλος. Η Καρολίν προσβλέπει στη συνεργασία μαζί σας στις επόμενες συναντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμος αντικαταστάτης είστε σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο στο όνομα τη Γκουε, όχι, ούτε έχουμε κάποιον από το ENF. Να δώσω λοιπόν το λόγο. Α, μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο ή κάποιος άλλος ευρωβουλευτής. Παρακαλώ. Αγαπητέ σκιώδη συγητά των σκιωδών Σιγητών, αγαπητέ Αλέν. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι κατά βάση να έχουμε ενσωματώσει όλες τις τροπολογίες των ομάδων που έχουν ε, λάβει το λόγο, άρα και του κυρίου Στόλογιαν, τις τροπολογίες, στα όσα είπε υπερβάνσο για τους σοσιαλιστές δημοκράτες. Δεν μπορώ παρά να πω ότι βεβαίως και υποστήριζω την πρότασή σου για ένα, τέτοιο, για ένα σεμινάριο, πλην όμως από τις ε, συζητήσεις μας εδώ αντελήφθην ότι στόχος ήταν να έχουμε μια πιο θεσμοθετημένη προσέγγιση και το είδαμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λάβαμε την πληροφορία ότι ε, υπάρχει περίπτωση τα κράτη-μέλη να το δεχθούν αυτό. Ένα γραφείο φυσκάλης Φερρυπίν που θα ήταν το κέντρο συντονισμού συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών δεν φαίνεται να θέλουν να το δεχθούν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό δεν το έχω βάλει στην έκθεση. επίση. δεν βλέπω τροπολογία από πλευρά σα που να ζητεί κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό και το απευθύνω στου σοσιαλιστέ δημοκράτες, αν πράγματι σας ενδιαφέρει, παρακαλώ φέρτε το θέμα τη στη συνεδρίαση τη ε, Τρίτη. Πολύ ευχαριστώ να το δεχθώ. Πέραν αυτού, για την Άλντε. Τις προτάσεις σας τις έχουμε συμπεριλάβει στις ε, συμβαστικές πλην μίας που κρίνουμε ως ε, νομικά αδύνατες. Μας λέτε ότι έχετε προτεραιότητες, κατάλογο προτεραιότητων για, τον, ε, για το πρώτο επίπεδο, που μετά θα διορθώσουμε με κατεξοδότηση πράξη. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Αν έχουμε πρώτο επίπεδο, δεν γίνεται τροποποίηση με κατεξοδότηση πράξη. Ή αλλιώς έχουμε κατεξοδότηση πράξη, αλλά όπως είπα, αν είναι στο πρώτο, στο πρώτο επίπεδο, δεν μπορεί μια εξοδότηση πράξη να, τις, ε, να τροποποιήσει διατάξει. Πολύ ευχαριστώ όμως να το συστήσουμε αν θέλετε. Αλλά για να μην μακρηγορούμε. Ελπίζω να συνεχιστεί καλή συνεργασία. Και να φροντίσουμε να ενισχύσουμε την διαφάνεια του φυσικάλης αλλά και την ε, καθοδήγηση σε πολιτικούς όρους από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους πόρους που επίσης χρειάζεται να έχει και αξίζει να έχει γιατί έχει αποδείξει την ε, προσθεμένη του αξία. Καλώς ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και εσάς και τους άλλους σκιώδεις. 27 Νοεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ολοκληρώσαμε και το σημείο 8 και ξανακάνουμε διάλειμμα. και νομίζω θα αναλάβει η κυρία Μπερές την ε, Προεδρία από εδώ και μπρος. Και την ευχαριστώ για την ευγενή της καλοσύνη. Συνεχίζουμε σε μερικά λεπτά λοιπόν. Euh, Ευχαριστώ. Ε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε λοιπόν τι ε, εργασίε. Φτάνουμε στο σημείο 9, βάσει το οποίο θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση της Νίνα Γκίλα σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με του δείκτε αναφορά χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του δείκτε αναφορά θετικού ενητικού άνθρακα. Μελετάμε τώρα ε, τι ε, τροπολογίες. Ε, έχουμε την ένδυ και την Ήτρε ε, οι οποίες θα κάνουν γνωμοδοτήσεις. Αγαπητή Νίνα Γκίλ, έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε την άποψή σας για τις ε, τροπολογίες. Είναι 242 τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω όλους, σε όλους ε, περί πρόκειται. Η ιδέα είναι ε, να έχουμε κοινούς δείκτες ε, αναφοράς ε, για την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα και θέλουμε να εστιάσουμε στην προσπάθεια οι δείκτες αναφοράς να ευθυγραμμιστούν με τη Συμφωνία των Παρισίων και βεβαίως πρέπει να το κάνουμε βλέποντας προς το μέλλον και οπωσδήποτε να υπάρξει διασύνδεση με την πρόταση ταξινομίας. Αυτό που θέλουμε είναι να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα τομέα ε, να υπάρξει μια καλή ανάλυση ε, των δαπανών και των τελών και βεβαίως αυτή η ανάλυση να είναι διαφανής καθώς επίσης να μελετήσουμε τον αντίκτυπο αυτού του κανονισμού όσον αφορά ε, τα οικονομικά είτε ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις και τη συμφωνία των Παρισίων. 240 είναι οι τροπολογίες από τους σκιώδεις στην ουσία αλλά και από μερικούς άλλους συναδέλφους. Ε, θα μπορούσα να, τους, να χωρίσω τις τροπολογίες σε τέσσερις ομάδες ε, τις οποίες έχουμε συζητήσει ως, εισηγη... ως σκιώδης. Πρώτον, ε, το όνομα αυτό, low carbon benchmarks κτλ. Ο τίτλος δεν υπάρχει συμφωνημένη συνένεση σχετικά με αυτούς τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ε, σε συνδυασμό και συνάρτηση με τα όσα αυτή η πρόταση προσπαθεί να επιτύχει. Θέλουμε όνομα και ορισμός να είναι σαφή έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα παρανόησης από πλευράς επενδυτών. Από την άλλη πλευρά βέβαια θέλουμε ε, τα οικονομικά και η βιωσιμότητα ε, να προωθηθούν ισομερώς. Πιστεύω ότι υπάρχουν ε, ε, στις 92 τροπολογίες που αφορούν το θέμα πολλές ε, προτάσεις. Από το climate transition, άλλη πρόταση θετική δείκτες αναφοράς, περιβαλλοντική δείκτες αναφοράς και Paris Benchmark. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα βέβαια είναι να κυκλοφορήσουμε έναν ε, συμβιβασμό στους συναδέλφους έτσι ώστε να δούμε αν και κατά πόσον μπορούν να ε, συμφωνήσουν. Και θα δούμε πώς θα πάει η συζήτηση την Τετάρτη. Δεύτερη μεγάλη ομάδα τροπολογιών, 25 συγκεκριμένα, αφορούν την ε, Κομισιόν και τις κατεξουσιοδότηση πράξης ξεκινούμε από διαγραφή οποιασδήποτε κατεξουσιώδηση πράξη από δράση κομισιών. Πολλή συζήτηση βέβαια έγινε μεταξύ του επίπεδου 1 και του επίπεδου 2, level 1, level 2. Έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες που θα κυκλοφορήσουμε και για το σημείο αυτό για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο το level 1, χωρίς να γίνουμε όμως και πολύ εξαντλητικοί και αναλυτικοί. Υπάρχει μια τρίτη ομάδα 50 τροπολογιών που αφορούν τα παραρτήματα. Και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα εμπλεκεί η Κομισιόν. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της, Ε, θα ακολουθήσουμε ένα μοντέλο αδειοδότησης, ας πούμε. Υπάρχουν διάφορες ε, μεθοδολογίες. Υπάρχει μάλιστα και μία πρόταση ο τομέας, η βιομηχανία να αποφασίσει μια και διαθέτει τεχνογνωσία για το θέμα αυτό. Τέλος, υπάρχει μία ομάδα που αφορά την ε, επέκταση της μεταβατικής περίοδου για σημαντικά, ε, σημαντικούς δείκτες αναφορές. Ε, τρεις τροπολογίες πάνω στα θέματα αυτά. Δύο από το ΕΛΚ, από, τον, την σκιώδη συγγήτρια Αν Σαντέρ και από τον Μάρκος Φέμπερ, συντονιστή του ΕΛΚ, και μία τροπολογία από την Άλτε, από την Καρολίνα. Γνωρίζω ότι υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το τι συμβαίνει με το benchmark ε, και με τον κανονισμό για τους δείκτες αναφοράς. Όμως δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι η λύση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος ε, των, ε, των δικτών αναφοράς μπορεί να βρεθεί η λύση λέω, του προβλήματος σε αυτό το θέμα και σε αυτό το κείμενο. Γνωρίζω ότι υπήρξαν παρόμοιες τροπολογίες στην για το θέμα ε, και αναρωτιέμαι το θέμα, ε, υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι θα πρέπει το θέμα οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί εντός του φακέλου αυτού, στα πλαίσια του φακέλου αυτού. Εμείς ε, προσωπικά πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σωστό και θα αντιτίθετο μάλιστα και στην ε, καλύτερη νομοθέτηση που θέλουμε εμείς, αλλά βεβαίως είμαι ανοιχτή για ε, περαιτέρω συζήτηση και ενδεχόμενη εξέβρεση συμβιβασμού και για το σημείο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πω κάτι άλλο. Ε, και να σχολιάσω τίποτα άλλο. Θα περιμένω πρώτα να ακούσω του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Για το ΕΛΚ, από ό,τι φαίνεται, λέει η Πρόεδρο ο Αλέλα Μασούρ θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και κυρία ε, Σκιώδη Πρόεδρε και, κυρία, και κυρίους και κύριοι Σκιώδη των Σκιωδών κτλ. Όμως θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα είναι η 40η ε, επέτειος ε, του θανάτου του ε, Ζακ Μπρέλ, Βέλγου τραγουδοποιού, ο οποίος έγραψε τρομερά τραγούδια, ένα από τα οποία λέει ότι άφησέ με να γίνω η σκιά σου, η σκιά του χεριού σου, η σκιά της σκιά σου, η σκιά του σκυλιού σου. exprimer devant euh, le point de vue Selon elle, ce règlement doit permettre la Λοιπόν, ε, ε, ελάχιστες απαιτήσει ε, για αυτούς τους δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα. Αυτά είναι πάρα πολύ θετικά πράγματα, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές. Διότι λέμε ότι θα πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούν με τις... Συμφωνία των Παρισίων. Ε, αυτό που θέλουμε βεβαίω είναι να μειωθούν ε, τα αέρια θερμοκηπίου και δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να, ε, ε να, να διαβρύνουμε τρομερά το κείμενο έτσι ώστε να γίνει δυσανάγνωστο για του επενδυτέ. Η Κομισιόν, όπω υπενθύμησε και η συγκήτρια, ε, προβλέπει κάποιε προτάσει επίπεδου 2 που δεν θα πρέπει να αφορούν μονάχα τα τεχνικά στοιχεία και το αναφέρει και η κυρία Σαντέρα. Όταν αναφερόμαστε σε πολιτικά στοιχεία, ε, και θέματα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διαιτησία μεταξύ των συνομοθετών. Όσον αφορά δε την ε, μεθοδολογία των διαχειριστών θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία των κανόνων έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ε, χρηματοδοτική καινοτομία και γρήγορη προσαρμογή στι ταχύτατα τροποποιούμενε συνθήκε. Στο παράρτημα θέλουμε όντω ευελιξία, η συγγήτρια αναφέρθηκε και σε αυτό. Σήμερα κάποιοι ε, ε, ε, κάποιοι δείκτες αναφέρονται μονάχα σε τρίτες χώρες και εκεί βρίσκονται και τα, οι δείκτες αυτοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020 πράγμα που οδηγεί σε κίνδυνο χρηματοοικονομικής αποσταθεροποίησης. Επίσης και λόγω του μεγέθους των μέτρων επίπεδου 2 προβλήματος στο κείμενο αυτό η Άννα θεωρεί ότι ο κανονισμός ε, θα, θα πρέπει να εφαρμοστεί μονάχα όταν θα έχουν δημοσιευθεί όλα τα στοιχεία του επίπεδου 2. Επίσης θεωρεί απαραίτητο σε αυτή τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία να μην αποκλειστούν κάποιοι ε, τομείς ε, γιατί ο στόχος, ο γενικός στόχος είναι να προωθηθούν όλοι μαζί και επομένως ο de facto αποκλεισμός ορισμένων τομέων ε, στην ουσία θα αντιτίθετο ή σε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ECR, υπάρχει κάποιος, κανείς. Για τους φιλελεύθερους έχουμε εδώ την σκιώδη εισηγήτρια και της δίνουμε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκίλ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως έχω και προηγουμένως πει, καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύω στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πρότασης για ε, όρια και προδιαγραφές μιας ευρωπαϊκής μάρκας δηλαδή σήματος που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε νέες προδιαγραφές για τις εκπομπές και αυτό σημαίνει ότι η χρήση των οροσίμων αυτών για τις εκπομπές θα είναι καθαρά εκούσια. Να, το να καταστεί λοιπόν υποχρεωτική και να προσδοριστούν προδιαγραφές για κάθε επίπεδο, για κάθε ορόσημο χαμηλών εκπομπών δεν είναι επιθυμητό γιατί ε, περιέχει τους εξής κινδύνους. Πρώτον, θα είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος υπάγεται στο πεδίο της και πολύ δύσκολο να την ε, αγνοήσουν, αγνοήσει κανείς. Δεύτερον, κινδυνεύουμε είτε να επιβάλλουμε μια μεθοδολογία έτσι καθυστερώντας ή εμποδίζοντας την ε, καινοτομία στην αγορά και δεύτερον να επιτρέψουμε στην Επιτροπή ή κάποιους άλλους να ορίζουν ποια είναι τα κατάλληλα ορόσημα που έτσι θα σφετεριστούν το δικαίωμα, την υποχρέωση καλύτερα της επιμέλειας που ανήκει στον καταναλωτή. Γιατί βεβαίω ε, δεν ε, μπορεί να καθοδηγήσει το κεφάλαιο μια τέτοια επιλογή μόνο Αυτό θα εξαρτηθεί μόνο από, το, ε, τον ίδιο τον επενδυτή. Ευχαριστώ κυρία Σκοτ Κάτω. Ευχαριστώ Περβάνο, ευχαριστώ και την Νίνα για την πολύ επικοδομητική δουλειά που έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό μέχρι τώρα και είχαμε πολύ καλό κλίμα στις συναντήσεις των σκιωδών που ήδη έχει οργανώσει. Υπάρχει συμφωνία ότι οι ορισμοί καθώς και οι ονομασίες ε, των δύο ε, δικτών ε, αναφοράς θα πρέπει να αλλάξει. Θέλουμε να είμαστε ε, φιλόδοξοι όσον αφορά την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ε, θέλουμε όμως να αποφύγουμε να είμαστε και ιδιαίτερα διατακτικοί όσον αφορά αυτούς τους δείκτες αναφοράς. Θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα από τις μεθόδους για τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει εδώ η ηγετική θέση. Πολύ χαιρόμαστε που η πρόταση για ε, μεταβατικό δίκτυ έχει γίνει θετικά αποδεκτή και πιστεύουμε ότι ε, τα benchmarks ε, για χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν. Αυτό αρχικά θα αφορά πολύ λίγες επιχειρήσεις, ε, θα είναι όμως ε, ιδιαίτερα υπέρ των επενδυτών που θέλουν να επενδύσουν σε πραγματικά περιβαλλοντικές επιχειρήσεις ε, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος σε ψευδούς ταυτότητα. ταυτότητας. Από την άλλη, θα πρέπει να μπορεί να, να αποδείξει κανείς ότι είναι προσιλωμένος στην απαλλαγή από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα για τις περισσότερες επιχειρήσεις που δεν, είναι ήδη, που δεν έχουν ήδη οικολογικό προσανατολισμό και θα βοηθήσει αυτό ε, την αναχρηματοδότηση όταν θα θέλουν αυτές οι επιχειρήσεις να ξεφύγουν από την ε, η δική τους θέση ως περιβαλλοντικές εταιρείες και να ε, μπουν στο γενικό ρεύμα. Πρέπει να υπάρξει θετική και συνεισφορά στην ε, μείωση των ε, εκπομπών ε, και όχι απλά να αντισταθμίζονται οι αμαρτίες τους από κάποια περιβαλλοντικά μέτρα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ποιοτικούς δείχτες που όμως να μην πνίγουν την καινοτομία. Οι πάροχοι των δικτών αυτών θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώσουν στις μεθόδους τους τα τελευταία ευρήματα. Κάποια στοιχεία στην πρόταση είναι περιτά, διότι υπάρχει επικάλυψη με άλλα τμήματα της ε, οδηγίας ε, για ε, τους δείκτες αναφοράς και αυτή το, το περιττό λίπος, να το πω έτσι, θέλουμε να το περικόψουμε. Επίσης ε, υπάρχει προσπάθεια τροποποίησης σε κάποιο τμήματος των ε, οικονομικών δικτών αναφοράς ε, που δεν σχετίζονται όμως με τους δείκτες αναφοράς για, τον, για το διοξίδιο του άνθρακα. Καταλαβαίνουμε ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας θέλει να πετύχει τους δικούς του στόχους. Δεν πιστεύουμε όμως ότι οι δείκτε αυτοί έχουν θέσει στη συγκεκριμένη πρόταση. Ακούστηκε ότι οι τροπολογίες αυτές είναι απαραίτητες ε, για να αποφύγουμε ε, τις ε, οικονομικές αναταραχές, τους κλειδονισμούς, αλλά δεν υπάρχει καμιά απόδειξη γι' αυτό. Όπως βλέπετε έχουμε εύρια συμφωνία και πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εισηγήτρια θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην συζήτηση. Δεν έχουμε όμως εκπροσώπους των άλλων ομάδων. Η Κομισιόν είναι εδώ, αλλά δεν θέλει να εκφραστεί, άρα δεν της δίνω το λόγο. Αλλά, αλλά, θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, ΣΥΡΠΑ είναι και μετά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αρκετοί από τους ε, συναδέλφους μας έχουν ε, ασχοληθεί με την ταξονομία ε, το, την έκθεση για τα βιώσιμα οικονομικά. Γνωρίζουμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο κλίμα, διότι τελικά θα δημιουργήσουμε φούσκες και προβλήματα όπως είναι αυτό του φινικελαίου, διότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο σε άλλους ε, τομείς ε, πρώτων υλών περιβάλλοντος και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ε, ούτε το θέμα της ε, ε, διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι δείκτες αναφοράς να αντικατοπρίζουν όλα αυτά τα στοιχεία. θα πρέπει να ενσωματώνουν την αρχή της μη πρόκλησης βλάβης και του σεβασμού στο περιβάλλον. Πάντως νομίζω ότι γενικά μπορούμε να είμαστε κάπως θετικοί και ενώ δεν έχουμε το σκεπτικό του μαύρου καταλόγου, της μαύρης λίστας σε, κανένα τμήμα αυτής της νομοθεσίας, Φαίνεται να είναι εφικτή η εφαρμογή των κανόνων αυτών, ε, να μην είναι όμως ο πιο αποτελεσματικός ε, τρόπος. Ε, τα, οι δείχτες αναφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τον αρνητικό αντίκτυπο και αυτό είναι κάπως δύσκολο να γίνει. οι δείκτες αναφοράς ε, θα πρέπει να βασίζονται σε κάποιους ε, άλλους δείκτες ε, και αναφέρονται αυτοί σε έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου αναφέρεται στην νομοθεσία για την κοινοποίηση πληροφοριών και τώρα αντικατοπτρίζεται και στην πρόταση για την ταξονομία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην πρόταση για τους δείκτες ε, αναφοράς ε, για τις ε, χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο στη βιοπικιλότητα, στο κλίμα. Όταν όμως γίνεται ο υπολογισμός, ο υπολογισμός θα πρέπει να βασίζεται στους εναρμονισμένους δείκτες που θα εκπονηθούν και με βάση την ανάλυση του κύκλου ζωής, ώστε να μην έχουμε διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού σε άλλους τομείς ή στις διάφορες νομοθεσίες. Αν χρησιμοποιήσει κανεί ε, τέτοιου δείκτε, ε, το πρόβλημα είναι ότι λέμε ωραία, έχουμε πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα, ε, δεν έχουμε ζημιά κοινωνική. διότι αναφέρθηκε η μειονεκτηματα οσον αφορα τη βιοποικιλοτητα θετικο η αρνητικο αντικτυπο στο κλιμα δεν εχουμε ζημια κοινωνικη διοτι αναφερθηκε η υποθεση του φινικελαίου, όπου μπορεί να έχουμε θετικό αντίκτυπο σε ένα τομέα, αλλά πολύ αρνητικό σε άλλο. Εάν εφαρμόσουμε την ανάλυση του κύκλου ζωής, εάν ε, εισάγει κανείς φινικέλο, για παράδειγμα, από άλλα μέρη του κόσμου, μπορεί να έχουμε πολύ αρνητικό οικολογικό αποτύπωμα τελικά. Και έτσι να μην μπορούμε να θεωρήσουμε θετικό έναν δίκτυ που ενθαρρύνει τέτοιου είδους δραστηριότητες. ένα από τα βασικά βήματα όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων ε, και, την, ε, και το μετριασμό της ε, αλλαγής του κλίματος. Πρόκειται εδώ για ένα σημαντικό βήμα, γι' αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σωστά και θα χρειαστεί εναρμονισμένη προσέγγιση και όσον αφορά την ταξονομία και την κοινοποίηση πληροφοριών. Αυτό το σκεπτικό διέπει τις τροπολογίες μου και γι' αυτό ελπίζω να μπορέσετε να τι λάβετε υπόψη σας όταν ε, καταλήξετε σε συμβαστικές προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριο Στάν. Συμφωνώ κι εγώ ότι πρέπει να κοιτάμε και το κέρδος και τον πλανήτη και τον πολίτη και συμφωνούμε πιστεύω και σε ένα άλλο ζήτημα σαφές νομίζω με τις θέσεις που υθετήσαμε στη Ρήτρα για τη δέουσα επιμέλεια ότι το Κοινοβούλιο δεν θέλει να κολλήσει μόνο σε μια πράσινη προσέγγιση αλλά ότι θέλουμε να ενισχύσουμε με τις ε, με τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, το πρόγραμμα δράση να είναι σαφές δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καινοτομία και δυναμικό υπάρχει αλλά πρέπει να απελευθερωθεί. Για τα ορόσημα. Το κείμενο από την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου των εμπειρογνωμόνων έχει πει ότι είναι πολλές φορές παραπλανητικό το να υπάρχουν ορόσημα που τα παρακολουθούν οι πάντες. Και έχει δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και έχω ε, προβλέψει και συμφωνώ με τα όσα είπε η ΣΥΡΠΑ ότι πρέπει να ευθυγραμμιζόμαστε με τη Συμφωνία για το Κλίμα. Έτσι λοιπόν η τροπολογία μου προβλέπει σε τέσσερα χρόνια τα ορόσημα να έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρω με τη Συμφωνία των παρουσιών. Και αυτό μπορεί να είναι μία ε, πρόταση, αλλά το όνομα της δικής μου της τροπολογίας ήταν να ευθυγραμμιστεί το ESG στην, ε, στον τρόπο λήψη αποφάσεων για τις επενδύσεις. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση της Νίνα Τζέιλ, ότι δηλαδή μόνο, σύμφωνες με την, μόνο σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων δεδομένα μπορούν να ενσωματώνονται στα κρίσιμα ορόσημα. Δηλαδή, όλα τα ορόσημα πρέπει να προσαρμόζονται και να ευθυγραμμίζονται με τη Συμφωνία των Παρισιών, αλλά τα κρίσιμα πρέπει να είναι και υποχρεωτικά ευθυγραμμισμένα. και νομίζω έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ενσωμάτωση όλων των μελημάτων του ESG στις ε, προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Θέλω και εγώ να λάβω το λόγο. Ναι, ορόσημα για τον άνθρακα. Από την άλλη όμως έχουμε και όλες τις συζητήσεις της ομάδας ψηλού επίπεδου με τη δυνατότητα διεύρυνσης του φάσματος για να συμπεριληφθούν και όλες οι πτυχές ε, ESG, περιβάλλον, κοινωνικά και τα λοιπά. Και όταν είχαμε τη συζήτηση με τον Τίμαν, άλλωστε το είχαμε επισημάνει αυτό, ότι αν ε, περιορίζουμε υπερβολικά ε, τις επιλογές μας ως προς τον άνθρακα θα κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ευκαιρία σημαντική. Ωστόσο εδώ έχουμε μια στρατηγική που μπορεί να αποτελέσει και τον κινητήριο μοχλό για να πούμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεύτερον, εάν κοιτάξουμε όχι μόνο το τεχνικό στοιχείο της αναθεώρησης των δικτών, ή να το πω αλλιώς, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί προσπαθούμε να διαρρήξουμε την απομόνωση των δύο σφαιρών που δεν συνομιλούσαν αφενός μεν χρηματοδότες ε, κεφάλαιο αφετέρου ε, περιβάλλον, περιβαλλοντική υποστήριξη κτλ. Και εδώ μπορούμε νομίζω να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα μελήματα περιβάλλον πρώτα αρχικά και μετά τα SG. Ε, που μπορούν βεβαίως να επιτρέψουν σε μια επιχείρηση, αλλά όχι μόνο να προβάλλεται ως ε, ευαίσθητο για το περιβάλλον ή μόνο για τα θέματα που αφορούν τον πολίτη, ε, πρέπει να καλύπτει όλα τα, όλους τους στόχους, όλα τα μελήματα. χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εγώ θα έλεγα να μην αναβάλουμε επαόριστον όλες αυτές τις προτάσεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε μέσα το κάνουμε. Ας μην ε, ε, παρασυρθούμε στην απέτηση να έχουμε πρώτα την ε, ονοματολογία ολοκληρωμένη για να προχωρήσουμε γιατί κατά πάσα πιθανότητα και βλέπω και τη δική σας ε, αντίδραση, από τη δική σας αντίδραση και, το, τα πρόσωπα σας θα είναι δύσκολο να το ολοκληρώσουμε στην τρέχουσα θητεία. Άρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε στο μέγιστο δυνατόν. Και από αυτά που είπε η συγγήτρια για τις τροπολογίες που είναι αυτό που θα λέγαμε στα γαλλικά νομοθετική υπότες, δηλαδή που θα μπορούσαμε να, να χρησιμοποιήσουμε για να ξανανοίξουμε την διαπραγμάτευση για το προηγούμενο κείμενο που αφορούσε τους δείκτες και τους, τα ορόσημα, τα κρίσιμα ορόσημα μάλιστα. Και εδώ έχω πράγματα που τα ξέρω και απ' έξω να σας τα πω, γιατί είναι τροπολογίες ακριβώς ταυτόσιμες με εκείνες που είχαν καταθέσει ακριβώς οι ίδιοι συντάκτες στο πλαίσιο της ε, αναθεώρησης των αρχών εποπτείας στο πλαίσιο της οποίας ο κανονισμός ή η η κρίσιμη, τα κρίσιμα ορόσημα ανοίγουν πάλι για την ε, αναθεώρηση από τις αρχές εποπτείας. Για να έχουμε λοιπόν συνεπιστάση εάν αποφασίσουμε ότι πρέπει να χειριστούμε το θέμα αυτό, που είναι και ζήτημα χρονοδιαγράμματος και υλοποίησης των κρίσιμων οροσίμων. Και όπου μας λένε οι υποπτικές αρχές, μα είναι περίπλοκα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν τα καταφέρνουμε, χρειαζόμαστε και χρόνο. Αυτή τη συζήτηση ας την αφήσουμε για να γίνει με την ευκαιρία της αναθεώρησης των αρχών εποπτείας ή όπου άρχισε να ανοίγει αυτός ο κανονισμός. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η θέση του Προέδρου μας, του Πρόεδρου της Επιτροπής. Η συγγήτρια, παρακαλώ για να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συνάδελφους για τα σχόλια. Ιδίως τους Σκιώδης που θα ξανασυναντήσω αυτήν την εβδομάδα. Για τους λοιπούς... Για να απαντήσω σε κάποια από τα μελήματά σας, μια και δεν θα είστε με, την, ε, με τους σκιώδεις όταν ε, έρθει η ώρα να τους δω, για την ε, Σύρπα και τον Πόρλο η αρχική μου πρόταση στο σχέδιο προτάσεως ιδιαίτερα έδινε έμφαση στην συμπερίληψη του S και του G, όχι μόνο του ε, δηλαδή όχι μόνο του περιβάλλοντος. Και το τονίζω αυτό άλλωστε στο σημείωμά μου ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τόσο επί ομάδα υψηλού επίπεδου. Τώρα, στο αν θα πρέπει κάποια ορόσημα ή όλα να είναι προγραμμισμένα. Η αρχική μου πρόταση ε, ανέφερε ότι έπρεπε να είναι όλα τα ορόσημα ευθυγραμμισμένα, αλλά η αντίδραση από όλους τους σκιώδεις συνολικά, συνολικά πλην ενός ίσως, ήταν ότι δεν μπορούμε να ειναι ολα τα οροσημα ευθυγραμμισμενα αλλα η αντιδραση απο ολους τους σκιωδη συνολικα συνολικα πλην ενος ισως ηταν οτι δεν μπορουμε να περασουμε τη λύση των, ε, της ευθυγράμμισης για όλα τα ορόσημα και ακούστηκε αυτό στην αίθουσα νομίζω. Η δεύτερη τροπολογία λοιπόν στόχο είχε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα κέριο ορόσημο που θα είναι αυτό που θα λέγαμε κρίσιμο ή σημαντικό ιδιαίτερα. Γιατί περιμένω ότι δεν θα εγκριθούν όλα από όλου. Γι' αυτό θέλω να γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Αλλά όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. και νομίζω Πολ το βλέπεις και εσύ στην ε, έκθεσή μου ότι προσπαθούμε όντως να εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση. Είναι σημαντικό αυτό για το Κοινοβούλιο και προσπαθούμε και στις συζητήσεις για τις συμβιστικές τροπολογίες να, να εξασφαλίσουμε ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό ως προς την άποψη αυτή. Βλέπα βέβαια και ανάμεικτες αντιδράσεις από τους συναδέλφους για την εισαγωγή ενός χρονοδιάγραμματος. Ε, αυτό νομίζω θα το δούμε, Πρόεδρε, στις ομάδες εργασίας. Και ξέρω ότι δεν ήθελα να σχολιάσει η Επιτροπή, αλλά θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για παρατηρήσεις που ακούστηκαν στην ομάδα εργασίας. για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των εκπομπών. και ένα από τα σχόλια είναι ότι είναι σε αυτές οι μέθοδοι και όσο πρέπει να εγκαταλειφθούν. Μπορεί η Επιτροπή τουλάχιστον αυτό να μου το σχολιάσει. Πόθεν προέρχονται αυτές οι μεθοδολογίες. Είναι κανείς εδώ να μας απαντήσει. Γιατί θα το χρειαστώ και την ε, συζήτηση που θα έχουμε την Τετάρτη. Παρακαλώ. Euh, est-ce que la άλλαξε γνώμη Επιτροπή, Σα ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σα. Όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα της μεθοδολογίας, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά, κάτι που συμπεριλαμβάνεται στην εντολή της τεχνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων που αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει τις εργασίες της και ένα από τα βασικά καθήκοντα της ομάδας αυτής είναι να καθορίσει την καλύτερη μεθοδολογία καθώς και να συλλέξει όσο γίνεται περισσότερα δεδομένα σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά και να συμπεριλάβει και αυτήν την διάσταση ε, στους δείκτες αναφοράς χαμηλών ε, ανθρακούχων εκπομπών. Συμπεριλαμβάνεται λοιπόν στη θητεία, στην εντολή συγγνώμη, της ομάδας αυτής το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ άψογα. Ευχαριστούμε και για αυτές τις διευκρινήσεις που είμαι σίγουρη ότι βοήθησαν και θα βοηθήσουν την εισηγήτρια στην προσπάθεια εξέβρεσης συμβιβαστικών ε, τροπολογιών. Ψηφοφορία θα λάβει η χώρα την 3η Δεκεμβρίου για το θέμα αυτό. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 10 της μερισίας διατάξεως. Πρόκειται για την έκθεση του Wolf Klintz ε, σχετικά με τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων από ό,τι καταλαβαίνω, ο συντονιστής της ε, ομάδας ε, Άλντε ε, θα παίξει το ρόλο του σκιώδου του εισηγητού και επομένως θα δώσω τον λόγο στον αγαπητό φίλο που θα λάβει αυτήν την παίξει αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως βλέπετε ο, Γουλφ ο Κλίντς Γουλφ δεν είναι εδώ ε, και επομένως θα μιλήσω βασιζόμενο σε κάποιες σημειώσει που μου είχε αφήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δυστυχώ δεν τα κατάφερα να είμαι ε, κοντά σα. και ε, έχω λοιπόν να δηλώσω ορισμένα πράγματα. Οι τροπολογίες ε, οι οποίες έχουν κατατεθεί ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση με την έκθεση, ε, ε, με το προσχέδιο έκθεσης και επομένως υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλών τροπολογιών. Επίσης μας λέει ο εισηγητής ότι έχουν προετοιμαστεί 7, σκιό, 7 συμβιβαστικές που έχουν σταλεί στους σκιώδεις. Θα συζητηθούν τούτη την Τετάρτη ε, και ε, προκύπτουν τρία στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Πρώτον, ο ορισμός, ε, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις του pre-marketing δεύτερον οι προϋποθέσεις αυτού του καθεστώτος και τρίτον ο καθορισμός των marketing activities. το ένα σημείο το οποίο μας απασχολεί είναι το μέλλον των BRIPS. Κατά την έννοια αυτοί, ΕΛΚ και ΣΥΑΡ έχουν υποβάλει κοινή τροπολογία για το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο είπε τώρα ότι θα συμφωνήσει με την πρόταση του Κοινοβουλίου. Επομένως, ερώτηση προς την Κομισιόν από πλευρά του Wolf Klintz βέβαια. Μπορεί ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να μας πει σήμερα σύντομα εάν δέχεται ε, η Κομισιόν αυτή την προτινόμενη λύση. Αυτή είναι η ερώτησή μου και ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για το ΕΛΚ. Ο Σκέδης συγητής είναι ο Μασούρ. Θα του δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ ε, πολύ. Αυτή τη φορά παίρνω τον λόγο σαν πραγματικός ε, σκιώδης. Θα ήθελα βέβαια να συγχαρώ τον εισηγητή για την σημαντική εργασία που έχει ολοκληρώσει και για τον τρόπο με τον οποίο ε, διαρκώς ζητούσε την άποψη και ενέπλεκε τους σκιώδης στην διαδικασία αυτή. Θα υπενθυμίσω εδώ όμως κάποια σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά. Όσον αφορά το pre-marketing, φαίνεται να προκύπτει ε, συμβιβας, συνένεση και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό έτσι ώστε το pre-marketing να θεωρηθεί ε, προϋπάρχον ε, ταμείο ε, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και σε άλλες χώρες όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και ε, ε, εγγύσεις όσον αφορά τα reverse solicitation και αυτό είναι πολύ θετικό. Παραμένει μία δυσκολία όσον αφορά την επέκταση και στο usage Κατά την δική μας άποψη, τα on usage ε, αφορούν την λιανική retail και επομένως δεν υπάρχει λόγος να μην διευκολυνθούν ε, και ε, τα euh, euh, euh, τα κεφάλαια αυτά και να αφορούν και τις πιο μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τον λόγο της ΕΣΜΑ. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα η δημιουργία ενός πορταλέσμα ε, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή ε, σχέση ανάμεσα ε, στις αρχές προορισμού και στις αρχές κίνησης και βεβαίως καλή συνεργασία με τις εθνικές αρχές και εάν πρέπει να ε, υπάρχει όλος αυτός ο συντονισμός θα ήταν θετικό ε, να περνάει μέσα από την ΕΣΜΑ λαμβάνοντα πάντα υπόψη και σεβόμενη, και τις αρχές του ε, νομοθετήματος προσπέκτους όσον αφορά τα τέλη. Συμφωνούμε με εξορθολογισμό των, του κόστους που θα είναι αιτιολογημένη και θα συνδέεται με μια ε, ε, διαδικασία πραγματικής επιτήρησης. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την, ε, την τροπολογία του Ryan που αφορά το MMF και υποστηρίζεται και από το ECR. Πιστεύω ότι είναι μια συζήτηση από την οποία έχουμε όλοι εξαιρετική, εξαιρετικές αναμνήσεις από τη συζήτηση, αλλά δεν θέλουμε να την ξανανοίξουμε ένα άλλο σημείο το οποίο αφορά ε, την ε, εξαίρεση των usage στο φάκελο Πρίψε. Κατανοώ ότι ο εισηγητής από ό,τι φαίνεται μετά από δικιά σας πρόταση είναι διατηθειμένος να οργανώσει συνάντηση με την Κομισιόν και βεβαίως εάν αυτή η συζήτηση πραγματοποιηθεί θα ήμουν ευτυχής να συμμετάσχω. Σοσιαλιστική ομάδα Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και να ε, επιβεβαιώσω ότι πράγματι λάβαμε και εμείς συμβαστικές τροπολογίες και θέλουμε και εμείς να βρούμε λύσεις ε, στο θέμα αυτό. Εμένα η βασική μου ανησυχία είναι η προστασία των επενδυτών. Μας ενδιαφέρει δηλαδή, το θέμα της κοινοποίησης. Φυσικά θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις διασυνοριακές δραστηριότητες και θα πρέπει να μπορεί κανείς ε, να ε, ε, εισέλθει και να αποχωρήσει από μια αγορά χωρίς περιπλοκές. Μας ενδιαφέρει όμως και η προστασία του επενδυτή και γι' αυτό προτείνω στις τροπολογίες μου να είναι δυνατή η αποχώρηση εφόσον ε, δεν έχει απομείνει κάποιος λιανικός επενδυτής στις αγορές αυτές. Εάν όμως υπάρχει οποιοδήποτε επενδυτής ε, στην αγορά υποδοχής θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς και να ενημερώνεται σωστά. Στο ίδιο πνεύμα θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι υπέρ των ανοιχτών αγορών ΟΣΕΚΑ στο θέμα αυτό, διότι ε, η ΟΣΕΚΑ είναι προϊόν λιανική. Εάν λοιπόν εισάγουμε αυτή την τροποποίηση, δεν ξέρω ποιε θα είναι οι συνέπειε. Δεν υπάρχει σχετική μελέτη αντικτύπου και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες ε, της πράξης αυτής ε, προτού κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίσης ε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουμε το θέμα του πολιετού σε δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν βλέπω να είναι κάτι τέτοιο χρήσιμο την παρούσα στιγμή. Και τέλος, έχω μπερδευτεί κάπως με τις διάφορες προτάσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, ε, τις σχέσεις δηλαδή ανάμεσα στις εθνικές αρχές. Ε, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να ενημερώνεται εκ των προτέρων η χώρα υποδοχής σε σχετικά με την πρόθεση ε, των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης. Μπορώ να δεχτώ οι εθνικές αρχές να λαμβάνουν εκ των υστέρων τις πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να ενημερώνονται οι αρχές εκ των προτέρων. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εθνικές αρχές ε, και ε, τον ΕΣΜΑ, Πιστεύω ότι πρέπει να φροντίσουμε να διαβιβάζονται τα απαραίτητα δεδομένα. Δεν θα πρέπει όμως να πλημμυρίσουμε τις αρχές με υπερβολικά πολλά δεδομένα, διότι και αυτό δεν είναι χρήσιμο. Θα ήταν χρήσιμο ο ΕΣΜΑ να μπορέσει να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και πώς αυτές θα μπορέσουν να συμπληρωθούν. Επίσης προτείνω να γίνει προσαρμογή των πληροφοριών ε, και των επαφών ανάμεσα στις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές και του ΕΣΜΑ. Νομίζω πάντως ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ε, με, την ικανότητα του εισηγητή μας ε, θα φτάσουμε σύντομα σε συμβαστικές προτάσεις. Ο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να επικεντρωθώ στα βασικά στοιχεία. Γενικά συμμεριζόμαστε τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του εισηγητή καθώς και της πλειοψηφίας των Ευρωβουλευτών να ανοίξουμε τις αγορές υπό το φως της Ένωσης Κεφαλαιογορών ε, χωρίς να εισάγουμε περιτά εμπόδια στην μεταφορά κεφαλαίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή πράγματα που είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος ουσιαστικά. Πέρα από αυτό όμως, έχουμε ακόμα κάποια θεματάκια. Ε, οι συμβαστικές τροπολογίες ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι όσον αφορά την συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τις αγορές, πιστεύουμε ότι ε, θα είναι πιο κατάλληλο να έχουμε υποχρεωτική ρήτρα και όχι ε, προαιρετική, να έχουμε shell αντί για may. Όταν δηλαδή εισάγουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, να έχουμε υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε οι άνθρωποι να μην νιώσουν ότι η ισχυρότερη ε, ένωση κεφαλαιοχωρών οδηγεί σε, απώλεια, ε, του επίπεδου, σε μείωση του επίπεδου προστασίας του καταναλωτή. Χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε στη συμβαστική πρόταση του άρθρου 2 ότι αναφέρεται ο κίνδυνος και ε, η επιβράβευση και ότι οι κατευθυντήρες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της πρότασης αυτής Ε, έχει αναβαθμιστεί και τώρα πια μιλάμε για ATS. Ε Επίσης, Αναφέρεται ότι η εμπορική πρόθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ε, με πληροφορίες και θα πρέπει να γίνεται αναφορά των εθνικών και ευρωπαϊκών ένδικων μέσων. Έτσι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των συλλογικών επενδυτών. Και όσον αφορά τα θέματα πριν ε, τη διάθεση στην αγορά, πριν την εμπορική πρόθεση, αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βρει πολύ καλή ισορροπία και είμαστε υπέρ της διατήρησης της πρότασης ως έχει πρέπει να περιορίσουμε τις δράσεις πριν τη διάθεση στην αγορά στις προϋποθέσεις που αναφέρονται. Επίσης ε, χαίρομαι διότι η τροπολογία σας 135 σχετικά με την άτυπη ενημέρωση πριν τη διάθεση στην αγορά. Ε, αυτό είναι πολύ θετικό βήμα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι η αποδυνάμωση του κανονισμού για τις ε, χρηματικές αγορές ε, είναι κάτι που έχει υποστηριχθεί από τους συναδέλφους Hayes και Καμάλ από το ECR. Αυτό φαίνεται να είναι κακό γουστο αστείο. Χαίρομαι λοιπόν που οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες έχουν αντιδράσει και δεν δέχονται την εισαγωγή πιο αυστηρών κανόνων για τα σύναυς. Χαίρομαι που αυτή η πρόταση ουσιαστικά πέθανε πριν ε, εφαρμοστεί. Πρόκειται για πολύ καλή κίνηση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που στην συνάντηση των Σκιωδών αυτή την εβδομάδα θα συναντηθούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με ε, τα κρυψ και το usage, τα, ε, τους οσεκά δηλαδή, που είναι ε, πολύ χρήσιμο διότι αν περιμένουμε ακόμη περισσότερα, σχετικά με το PRIPS, αυτό δηλαδή το βασικό ενημερωτικό στοιχείο, θα διακυβευτεί το σύνολο της πρότασης. Από την άλλη, αυτό το ενημερωτικό έγγραφο είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λειτουργήσει καλά και γι' αυτό περιμένω να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι πράγματι θα λειτουργήσει σωστά. Θα πρέπει κατά τα άλλα όμως να μείνουμε στα όσα ψηφίσαμε και να έχουμε αυτό το έγγραφο ως βασικό και καθολικό εργαλείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ε, έχουμε εκπρόσωπο της ΓΚΟΕ, άλλοι εκπρόσωποι ε, κομμάτων ο σκιώδες δεν υπάρχουν. Θα δώσω το λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πριν από αυτό ίσως και εγώ να πω δύο λόγια. Επανερχόμενοι σε δύο θέματα. Το πρώτο για το νομισματικό ταμείο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ξανα ε, μπήκε στο θέμα. Νομίζω ότι η θέση των μεγάλων ομάδων ε, και από ό,τι καταλαβαίνω και των πρασίνων ε, είναι συγκεκριμένη. Δεν άκουσα τη γνώμη του εισηγητού, αλλά ίσως ο σκιώδης του εισηγητού να μας πει δύο λόγια και γι' αυτό. Πιστεύω ότι ως νομοθετική πρακτική αυτό δεν θα ήταν καθόλου καλό, γιατί όλοι θυμόμαστε τις συζητήσεις που είχαμε και με την ΕΣΜΑ και με την ε, Κομισιόν όσον αφορά την αναγνώριση του δημοσίου ε, χαρακτήρα της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν ε, που μας είπε τι συμβαίνει με το θέμα αυτό και με το φάκελο αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει πλήρως να ακολουθήσουμε τον νομοθέτη ε, να μην λάβουμε υπόψη μας αυτούς ε, τους νομοθετικούς ε, αναβάτες και υπείς. Όσον αφορά το πρίψ τώρα και την την, ε, στο με τον, ε, την νομοθεσία βέμα. Στο επίπεδο 1 είχαμε πει ότι θα υπάρχει πρώτα μια αξιολόγηση και μετά να δούμε την εφαρμογή ε, στα, στο τμήμα των OPCVM. Ε, VM. Κάποιοι σήμερα βασίζονται στην καθυστερημένη θέση ισχύ των PRIPS έτσι ώστε να ε, καθυστερήσουν όλη τη διαδικασία. Όμως σημειώνω ότι σε μια χώρα όπου υπήρχε ισχύρος λόγος για την ε, μετάθεση της θέσης ισχύ των πρίψε, λαμβάνω σήμερα επιστολές από καταναλωτές και από οργανώσεις ε, καταναλωτών ε, που εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την μη εφαρμογή των πρίψ στα OPCVM. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση. Θα είναι οπωσδήποτε ορθολογική και σίγουρα όχι ιδεώδης. Εγώ όμως θα ήθελα να πάμε προς μια λύση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν θα πρέπει να είναι στο πόδι φυσικά, γιατί δεν υπάρχει και πολιτική συνένεση για να ζητήσουμε στις εποπτικές αρχές να κάνουν εργασία επίπεδου 2 από τώρα μέχρι το τέλος της θητείας. Ωστόσο, πιστεύω ότι το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Θα το συζητήσουμε με τον εισηγητή και την Κομισιόν. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να ε, ε, καθυστερήσει. Ε, θα ήθελα να ε, ζητήσω την Κομισιόν να πάρει το λόγο, χωρίς όμως ε, να αναφερθεί λεπτομερό σε όλα αυτά τα στοιχεία και τα λοιπά. Γιατί θα συναντηθούν και οι σκιώδες σε, σε μερικές μέρες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που σας απασχολεί και ευχαριστώ που ασχολείστε με αυτό. Κατά την άποψη της Κομισιόν, η έννοια του pre-marketing θα πρέπει να συνδυαστεί με, την, ε, με, τις ε, εγγύσεις ε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η σωστή προδιάθεση για τις αρχές επιτήρησης. Όσον αφορά την denotification, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είναι εναρρωσμένες οι προϋποθέσεις, όχι ε, να ληφθούν, να τεθούν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δυναμητήσουν την κατάσταση. Επίσης μπορούν να υπάρξουν και κάποιες εθνικές διατάξεις με την προϋπόθεση ότι διευκολύνουν την κατάσταση. Όπως αναφέρθηκε, η Κομισιόν δεν υποστηρίζει την τροπολογία σχετικά με τον ε, ε, την αντίστροφη ε, ροή. Και αυτό ε, αναφέρεται άλλωστε και στον κανονισμό που αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Άλλωστε μια τέτοια διαδικασία θα ήταν και θα ερχόταν και σε αντίθεση με την ultimate goal Σχετικά με την προληπτική διαχείριση και έλεγχο, ε, το ε, BRIPS μπορεί να ληφθεί υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι ε, μπορεί να είναι διπλό βάρος εάν δεν προσέξουμε και δεν θέλουμε. Θέλουμε να αποφύγουμε την διπλή επιβάρυνση βεβαίως. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο ακόμα χρόνια πάντως και μπορούμε να δεχτούμε την προδυνόμενη λύση λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί ένα βήμα προς ε, την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση όπου όλοι θα ξέρουν ακριβώς το ρόλο τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο φτάσαμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτητα ε, στις περαιτέρω αλλαγές ε, στο επίπεδο 2. Επίσης, μπορούμε να φτάσουμε και σε μία ενδεχόμενη αναθεώρηση των πρίψε, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Το δεχόμαστε, αλλά θα πρέπει να το δούμε στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης. Είναι σημαντικό τώρα να έχουμε τα πρίψε ε, και όσο γίνεται με ευρύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ξαναδίνω. Είναι εδώ ο σκιώδη του εισηγητού. Όχι. Θα μεταφέρθει πιστά στο Wolf Klintz το σύνολο των διαμυφθέντων. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Για την διατύπωση των τελευταίων συμβαστικών προτάσεων. Μακροσκελής φαίνεται ότι θα είναι η ψηφοφορία στις 3 Δεκεμβρίου. Ολοκληρώσαμε τα σημεία 10 και 11 λοιπόν. Σημείο 11. Ετήσια έκθεση Τραπεζικής Ένωσης 2018. Νίλ Στόρβαλς και Διλ. Παίρνετε το λόγο παρακαλώ για τις 186 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, 180 και ήταν οι τροπολογίες μας. Πολλές φορούσαν λογική σκέψεις βέβαια. Προσπαθούμε να τις ε, διευκρινίσουμε. Πρόβλημά μου, όχι δικό σας βέβαια, είναι το πώς θα διατηρήσω τη συνοχή και τη συντομία της έκθεσης. Ακόμα και για δημοσιογράφο, όπως εγώ, δύσκολο φαίνεται να είναι. Επικοδομητικές επιτοπλίστων των τροπολογίες. Δεν βλέπουμε δηλαδή να διασκοπίζονται προς απίστευτες και απίθανες κατευθύνσεις οι τροπολογίες. Αλλά όταν συντάσω τις συμβαστικές τροπολογίες, προσπαθώ να λαμβάνω υπόψη στο δυνατόν περισσότερες από τις τροπολογίες των συναδέλφων. Πράγμα δύσκολο μερικές φορές, γιατί υπάρχουν ομάδες που ακολουθούν τελείως αντιδιαμετρικές κατευθύνσεις. Και έτσι αυτό δεν είναι, δύσκολο, δεν είναι εύκολο να το συνδυάσουμε. Προσπαθούμε να βρούμε όμως μία διατύπωση που να καλύπτει και τις δύο μεγάλες ομάδες. Ε, και να διατηρήσουμε στο δυνατόν τη συνοχή του κειμένου. Ταυτόχρονα έχουμε προτάσεις που βγαίνουν σε διαφορετικά σημεία του κειμένου με τις τροπολογίες και προσπαθούμε να τα ενοποιήσουμε σε ένα σημείο για να μην έχουμε επανάληψη των ίδιων ε, ευχολογίων σε διαφορετικά άρθρα. Καλό λοιπόν τους ε, σκιώδης ηγητές να διατηρήσουν την επικοδομητική στάση που είχαμε και στο παρελθόν, στην πορεία μας μέχρι τώρα και να κοιτάξουμε μαζί τις συμβαστικές τροπολογίες και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να λάβω υπόψη όλες τις τροπολογίες και τις παρατηρήσεις σας. Ταυτόχρονα όμως ζητώ να τηρήσουμε και μια λογική γραμμή, αναλογική γραμμή, να μην ε, επεκταθούμε σε υπερβολικά πολλές ε, τροποποιήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, τροπολογίες. Βλέπω γενική υποστήριξη στην έκθεση και θα κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις σε επικοδομητικό πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουν εξηγήσει, θα, θα εξηγήσουν πιστεύω και οι συνάδελφοι τις προτεραιότητες τους. Ο Τόμας Μάν, σκιώδης από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ περβός και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Τόρβαλτς, πολύ καλή έκθεσή του και οι ιδέες του που μας ε, επανέλαβε και σήμερα η κύρια ιδέα πάνω απ' όλα να είναι όσο δυνατόν συνεκτικό το κείμενο και να μην επαναλαμβάνει διαρκώς τα ίδια πράγματα νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και στη συνεδρία των σκιωδών με αυτή την επικοδομητική στάση. Ε, εκ μέρους του ΕΛΚ αλλά και προσωπικά μπορώ και εγώ να εκφράσω την υποστήριξή μου σε πολλές από τις προτάσεις. Πάνω απ' όλα η Τραπεζική Ένωση να παραμείνει και να ενισχυθεί στη σταθερότητά της, ε, να εξασφαλίσουμε ισότιμες ε, συνθήκες για την εσωτερική αγορά και βεβαίως για τις τράπεζες έχει πολύ μεγάλη σημασία το κόστος, ιδιαίτερα για τις μικρότερες, ε, το κόστος που θα τις επιβαρύνει να μην ενισχυθεί σημαντικά. Γιατί βέβαια κινδυνεύει και η δυνατότητα προσφοράς χρηματοδότησης. Εμείς από το ΕΛΚ ιδιαίτερως ανησυχούμε για την διαφύλαξη, μεριμνούμε για την διαφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας που νομίζω ότι ήδη μας έχει ε, εξασφαλίσει η έκθεση. Η Τραπεζική Ένωση είναι ένα σαφής στόχος, μπορεί να έχουμε ε, διαφορετικές προσεγγίσεις και διαμετρικά αντίθετες για το έντις, ε, για, την, για τα αποθετήρια. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα βεβαίως τραπεζικά στις χώρες μέλη και πιστεύω ότι ε, καταγράφονται ικανοποιητικά στις ε, τροπολογίες που έχουμε δει. Χαίρομαι που και οι δικές μου αντικατοπτρίζονται στις συμβαστικές. Επίσης ε, πρέπει να διαφυλάξουμε την ποικιλία γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με την με τον πλούτο του τραπεζικού μας και του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μόνο σύστημα ή ένα μόνο τύπο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Χρειάζεται αυτή η διαφοροποίηση. Επίσης, υπάρχουν διάφορες διατάξεις περί αξιών που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Παραδείγμα, η πρόταση Επιτροπή για την ενίσχυση του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είναι ευπρόσδεκτη. Είναι κάτι το οποίο και ο πολίτη επιθυμεί και περιμένει. Δεν θέλει να οπισθοδρομήσουμε ε, σε μια κατάσταση όπου θα αποδειχθεί ότι κάποιες τράπεζες έκαναν αποτυχημένες επιλογές και κινδυνεύουν να καταστραφούν. Θέλουμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο ασφαλή κατάσταση στον τραπεζικό τομέα. Επίσης τα κράτη-μέλη πρέπει να περιγράψουν ε, το πρόβλημα σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η δε, το δε ζήτημα της, ε, του περιορισμού των μη, εξο, των εξυπηρετουμένων δανείων ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει τα κράτη-μέλη να επιληφθούν και πάνω απ' όλα να μην κάνουν τίποτα που να οδηγήσει σε χαλάρωση αυτού του συστήματος ε, της ενίσχυσης της ευρωστίας των τραπεζών. Οπωσδήποτε την Τετάρτη στην Επιτροπή, στη συνάντηση των σκιωδών θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό μια έκθεση πρωτοβουλίας με πολύ, καλά, με πολύ θετικά χαρακτηριστικά. Γιατί είναι απαραίτητο κάποια στοιχεία τα οποία βλέπουμε δυστυχώς να αναπτύσσονται σε κράτη-μέλη και μάλιστα δεν έχουν κάλυψη καμία να τα αντιμετωπίσουμε με τρόπο αποτελεσματικό και ε, με την επικοινωνία τη σωστή προς τον πολίτη εν ώψη και των ευρωεκλογών αλλά και γιατί ο πολίτης χρειάζεται αυτές τις απαντήσεις από πλευράς μας. Η Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σκιώδης ηγητής, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την εργασία του, διότι ε, προετοίμασε μια πολύ λογική και ισορροπημένη αρχική έκθεση. Ε, και τελείως ο αριθμό των τροπολογιών, που δεν ήταν και τόσες πολλές, κατέδειξε ότι παρότι υπήρχαν διαφορές, το αρχικό κείμενο είχε σωστό προσανατολισμό. Είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ορισμένες από τις συμβιβαλιστικές συμβιβαστικές τροπολογίες που προετοίμασε ο εισηγητής με τους ε, ε, σκιώτες. Υπάρχουν βεβαίως ακόμα και κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να βελτιώσουμε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βάλουμε την έκθεση αυτή ε, σε ένα σωστό πλαίσιο, γιατί ναι, είναι νομοθετικού περιεχομένου, έκθεση, ε, αλλά απαραίτητη, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για την Τραπεζική Ένωση, το πρώτο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει, η Τραπεζική Ένωση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ναι, έχουμε κοινό επόπτη, ε, κοινό ε, ταμείο εξυγίανσης, αλλά ακόμα δεν πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στοιχείο της ε, ε, Ευρωζώνης και κάθε φορά που και μια που θα συζητήσουμε για την Τραπεζική Ένωση είναι απαραίτητο το πρώτο που θα μας απασχολήσει στα πλαίσια της ε, Τραπεζικής Ένωσης είναι να δούμε εάν από καθαρά θεσμική ε, άποψη ακόμα χρειάζονται πολλά να γίνουν. Ίσως στο μέλλον όταν θα ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση ε, θα συζητήσουμε εάν λειτουργεί καλά, εάν λειτουργεί άσχημα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Τραπεζικής Ένωσης. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα θεσμικό πλαίσιο πλήρες για το σύνολο της Τραπεζικής Ένωσης. Επίσης, σημαντικό είναι να πούμε ότι για μια έκθεση ε, για την Τραπεζική Ένωση δεν θα ήταν σωστό να πούμε πώς θα εφαρμοστεί το banking package και τα λοιπά όλα αυτά τα οποία λειτουργούν εντός της ε, Τραπεζικής Ενώσεως χωρίς όμως να λέμε ε, σαφώς ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αυτή η Τραπεζική Ένωση και ότι οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ε, έναν μηχανισμό για τις καταθέσεις και ένα backstop για το σύνολο της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό πρέπει να είναι κεντρικό στοιχείο όλων των σχετικών εκθέσεων μέχρι ότου ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κεντρικό στοιχείο αφορά ε, τη λειτουργία, όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές τροπολογίες όπου γίνεται λόγος ε, για, τις, ε, για τους κινδύνους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Στο banking package ελπίζουμε ότι σε τριμερή διάλογο θα επιτύχουμε συμφωνία όσον ούπο, αλλά γίνεται και αναφορά στον νέο κανονισμό για τα MPRs. Είναι σημαντικό να δούμε αν θα συζητήσουμε, αν θα επιμείνουμε στην ανάγκη μείωσης των κινδύνων που συνδέονται ε, με τα MPLs, τα κόκκινα δάνεια και επίσης να δούμε τι γίνεται με τα ενεργητικά δευτέρου και τρίτου επίπεδου, επίσης ε, και με, τις, ε, με την χρήση των εσωτερικών μοντέλων που πολλές φορές αναμειγνύονται στον υπολογισμό ε, των ιδίων κεφαλαίων. Να δούμε λοιπόν όλα τα στοιχεία αυτά, αλλά πιστεύω ότι κυριότερο είναι να ε, ε, ασχοληθούμε και με τους κινδύνους ε, που σχετίζονται με το επίπεδο 2 και το επίπεδο 3 και να δούμε και τους επιπλέον κινδύνους του της Τραπεζικής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναφορά στην ολοκλήρωση το κλείσιμο της Τραπεζικής Ένωσης ασχέτως από ε, τους υπολογισμούς που κάνουμε εμείς για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η εγγύηση, η ασφάλεια των καταθέσεων κλπ το βέβαιο είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση των καταθέσεων επί τη βάση της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, και επιμένω ανάγκη να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τα διάφορα στοιχεία ενεργητικού χωρίς κινδύνους. Ε, βεβαίως το δημόσιο χρέο είναι κάτι τελείως ε, διαφορετικό ε, και θα πρέπει να βασίζεται σε ε, συμφωνίε συμφωνίες ε, και οπωσδήποτε να διέπεται από τις συμφωνίες της Βασιλείας και εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε αναθεώρηση που θα αλλάξει ε, την κατάσταση των, ε, των εθνικών, του εθνικού δημοσίου χρέους οπωσδήποτε θα πρέπει να συνδεθεί με τα ε, ενεργητικά χωρίς κινδύνους επί του συνόλου της Ευρωζώνης. Γι' αυτό το Sovereign Bond Bank Securities μας βρίσκουν σύμφωνους γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνουν την δυνατότητα συζήτησης για να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε ε, να αντιμετωπίσουμε την προληπτική εμπλοκή του δημόσιου χρέους βάσει των αρχών της Βασιλείας και ε, κυρίως για την Ευρωζώνη. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε ένα καλό αρχικό έγγραφο, μια καλή αρχική ε, έκθεση. Οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, και αυτό διαφαίνεται και από τις τροπολογίες. Ωστόσο, ε, πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε στην Επιτροπή εδώ και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ECR εκπρόσωπος. Για τους πρασίνους δεν βλέπω εδώ τον Ράλφο ε, Λάμπερ. Δεν έχω τίποτα που να θυμίζει πράσινο βουλευτή εδώ. Για το FDD επίσης δεν υπάρχει κανένας. Και για το ΙΕΝΕΦ επίσης δεν υπάρχει κανένας. Άρα, πριν ξαναδώσω τον λόγο, ε, να ρωτήσω εάν θέλει κανείς να πάρει το λόγο, έστω και αν δεν είναι αρμόδιος, όχι και επομένως δύο σημεία τα οποία αναφέρθηκαν και από άλλους συναδέλφους και τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον όσον αφορά ε, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τη μετατροπή του. Εγώ ε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, ε, βγάλουμε αυτήν την κακή ε, συνήθεια που έχουμε να ονομάζουμε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο την διάδοχο κατάσταση του EMS, του Μηχανισμού Σταθερότητας. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι έτσι ώστε να μην ε, συμφωνήσουμε με αυτήν την ονομασία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, Euh, de ne pas faire référence au mécanisme. Ε, πιστεύω ότι άσχετα από το, τα οσα δηλώνω το δηλώνονται δεξιά-αριστερά και τα διαστήματα από επίσημα ή ανεπίσημα χείλη, ε, δεν υπάρχει λόγος να ονομαστεί νομισματικό ταμείο. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, πιστεύω ότι θα ήταν αρκετά επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο, να υπάρξει παρανόηση όσον αφορά την νομισματική αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νομισματική αρμοδιότητα ε, αφορά την ε, ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελεία και παύλα και αλλάζουμε παράγραφο. Έτσι έχουν οι συνθήκες τώρα και δεν νομίζω ότι προτείνεται και τροποποίηση των συνθήκων. Δεύτερος λόγος, και ίσως και πιο αμφιλεγόμενος, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι το να γίνει αναφορά σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είναι ε, να δίνουμε την εντύπωση ότι στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο θέλουμε να εισάγουμε ε, ένα αντίγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όμως εμείς δεν είμαστε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε η Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο αντίστοιχο. Εμείς ε, έχουμε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει το μονοπόλιο της ε, άσκησης πρωτοβουλειών και επομένως δεν μπορούμε απλώς να αντιγράψουμε και να μεταφέρουμε κάποια θεσμικά στοιχεία και επομένως εάν μόνο το όνομα μεταφέρουμε και αντιγράψουμε κινδυνεύουμε να ε, ε, ε, προκαλέσουμε σύγχυση καθόλου επιθυμητή. Και όσον αφορά τη λέξη «πι» που χρησιμοποίησε ο Τόμας Μάνα, γιατί είναι μια συζήτηση που πλέον γίνεται οριζόντια, δηλαδή σε κάθε ε, ε, ε, περίπτωση και σε κάθε συζήτηση ξαναβγαίνει στην επιφάνεια το θέμα αυτό. Ναι, εσείς λέτε πρέπει να διατηρήσουμε την πολυμορφία, αλλά υπάρχει και η πολυμορφία των κινδύνων και υπάρχει και το γεγονός ότι το κάθε μοντέλο έχει τους δικούς του κινδύνους και το θέμα της αναλογικότητας δεν μπορεί να εξαντλήσει την ιδέα, την αντίληψη του κινδύνου και επομένως όταν μιλάμε ε, για το θέμα αυτό δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε μονάχα στους ε, κινδύνους που διαπιστώνει η ε, εποπτική αρχή, δηλαδή όχι μονάχα αυτή την αναλογικότητα αλλά και την αναλογικότητα του κινδύνου που θα μπορούσε αυτό το μοντέλο να παρουσιάσει για ένα συγκεκριμένο σύνολο αγοράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντίληψη της αναλογικότητας γιατί διαφορετικά θα περάσουμε για τίποτα χαζούς που δεν σέβονται το σύνολο των μοντέλων και δεν ε, ε, λαμβάνουν υπόψη τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία ε, των διαφόρων μοντέλων. Μακρηγόρησα αλλά δεν υπήρχε κανένας άλλος να πάρει το λόγο, επομένως καλά έκανα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για τη δική σα την τοποθέτηση. Δεν ήταν καθόλου μικρό και αντίθετο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η ιστορία με το Διεθνές Συμβατικό Ταμείο είναι παλιά, από το 69, όταν ήρθε ο Βίλι Μπραντ να πει ότι μπορούσε η Γερμανία να προσφέρει το 20% των νομισματικών της αποθεμάτων σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Έκτοτε λοιπόν κυκλοφορεί αυτή η ιδέα. Και μερικές φορές φαίνεται να μας συναρπάζει για να προχωρήσουμε. Αλλά θα προσπαθήσω να μην παρασυρθώ σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομος. o Και νομίζω και το όνομά του μας υποχρεώνει να ε, πούμε ότι δεν θα συντάξουμε μυθιστόρημα με τίτλο «Der Totin Venedicht», ο θάνατος στη Βενετία, ούτε όμως και ο «Der Totin Brüssel», θάνατος στις Βρυξέλλες. Mm. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τους σπόρους εκείνους που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε μια αποδεκτική ικανοποιητική λύση. Ακόμα και αν είναι τα δύο μεγαλύτερα, οι δύο πολύ μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες αντίθετες, έχουν τελείως διαμετρικά αντίθετες ε, θέσεις. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. και εύχομαι καλή συνέχιση στη δουλειά μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας. Πολύ χαίρομαι αν μπόρεσα και εγώ να συμβάλλω κάτι θετικό στις εργασίες σας. Εξετάσαμε λοιπόν και 27 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία και να κανονίσουν και οι ομάδες την παρουσία τους και την εκπροσώπησή τους και μάλλον έτσι ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Για αύριο πιστεύω να βρείτε άλλο πρόεδρο. Χαίρετε, καλό βράδυ.